Kära ledamöter, gäster och deltagare. Jag är glad att hälsa välkomna till eftermiddagens gemensamma möte mellan... Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα το απόγευμα έχουμε αυτή την ε, κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ε, με την Επιτροπή Γυναικών. Αν δούμε λιγάκι την, ε, το, το πώς αποκαλείται η σημερινή απογευματινή συνεδρία, θα δούμε ότι αναφέρεται πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει και να προλάβει κυρίως την εμπορία ανθρώπων και τι θα γίνει τελικά με το μέλλον. Έχουμε λοιπόν ε, μπροστά μας μια, ένα πολύ ενδιαφέρον απόγευμα θα έλεγα και έχουμε όμως και ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο πρόγραμμα. Θα ακούσουμε τις ε, απόψεις ε, πολλών ε, προσκεκλημένων μας που έχουν πάρα πολλές καλές γνώσεις όσον αφορά στην εμπορία των ανθρώπων και όλοι αυτοί θα μας εξηγήσουν πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Εν είδη λοιπόν, επιτρέψτε μου εγώ να αναφέρω τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας εξηγήσω τη διαδικασία. Η πρόταση την οποία θα εξετάσουμε σήμερα είναι το κείμενο της ε, Επιτροπής της Κομισιόν της 29ης ε, Μαρτίου. Αυτό είναι ένα σχέδιο οδηγίας για να ενισχύσουμε την ε, πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων. Ε, πρόκειται για το έγγραφο υπαριθμών 95. Όσον αφορά τώρα τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, αυτά κατά κύριο λόγο είναι γυναίκες και κορίτσια. Κατόπιν τούτου το θέμα αυτό εμπίπτει και στις αρμοδιότητες ε, των γυναικών. Αρμόδια λοιπόν η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών όπως επίσης και η Επιτροπή Ισότητας των Δύο Κατόπιν τούτου, όσον αφορά ε, σε αυτήν την έκθεση της ε, Κομισιόν, με βάση ε, το άρθρο 51 του κανονισμού, συνεργαζόμαστε για το θέμα αυτό. Κατόπιν τούτου το σεμινάριο, το απογευματινό, είναι κοινό και θα ήθελα να μου επιτρέπετε να ξεκινήσω παρουσιάζοντάς σας τους προσκεκλημένους. Έχουμε την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η οποία και θα αναλάβει ε, τον συντονισμό του δεύτερου τμήματος της συζήτησης. Έχουμε λοιπόν δύο εισηγητές, την Άννα Χέτ ε, από τους ε, σοσιαλδημοκράτες, σοσιαλιστές και δημοκράτες, η οποία εκπροσωπεί την Επιτροπή Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Πολιτικών Ελευθεριών και η επόμενη μιλήτρια που εκπροσωπεί την, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Οι δύο λοιπόν εισηγήτριες θα συμμετάσχουν ε, και στο, στην Προεδρία της ομάδας εργασίας. Να πω και κάτι άλλο. Έχουμε κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα. Ο κύριος Ρουής θα αντικατασταθεί από την κυρία Μαρτίνα Γκαρσία Αράντα και η Επιτροπή ε, θα εκπροσωπείται από τον κύριο Γιάκο Παρτίνσκι ο οποίος είναι και τμήματάρχης ε, αρμόδιος για θέματα οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, θα αντικαταστήσει τον κύριο Ράνχαρτ Πρίβεκ. Κυρία Λιντιέρ, που συμμετέχει στην Υποπιτροπή για, το, ε, για την Εμπορία Ανθρώπων στα, στο Συμβούλιο της Ευρώπης θα αντικαταστήσει την κυρία Λασεμπιάς. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους ομιλητές ε, να τηρήσουν ή δυνατόν το χρόνο που τους έχει διατεθεί. Και μετά θα διεξαχθεί συζήτηση. Στη συζήτηση ε, θα πρέπει όλοι οι συγητές να περιοριστούν στα δύο λεπτά. Οι ε, βουλευτές προηγούνται των υπολείπων όταν ε, θα φτάσουμε στις ερωταπαντήσεις. Τελειώνοντας λοιπόν, για άλλη μια φορά σας καλωσορίζουμε στο σεμινάριο και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών, η κυρία Άννα Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους θερμά σε αυτή την απογευματινή συνεδρίαση. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ακούσουμε πολλές και ενδιαφέρουσες απόψεις για το πώς μπορούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε την εμπορία ανθρώπων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Βρισκόμαστε στο 2010, όμως παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρώπη άνθρωποι που αγοράζονται και πολλούνται ως ε, σκλάβοι, παρότι η σκλαβιά καταργήθηκε πριν από 250 χρόνια. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί εξαναγκάζονται σε ε, επαιτία, ε, στην πορνεία και καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά. Αυτό είναι ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα στον κόσμο και παρόλα αυτά όμως ε, εξαπλώνεται το έγκλημα όλο και περισσότερο. Πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι εμείς κάνουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα αυτά. Γνωρίζουμε ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός ε, αποκλεισμό είναι ένα από τα βασικότερα αίτια που οδηγούν στην εμπορία ανθρώπων. Η ζήτηση ε, φτηνού εργατικού δυναμικού και σεξουαλικών διευκολύνσεων ε, επιδεινώνει το πρόβλημα. Άρα δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να αφορά όλους αυτούς τους τομείς. Εδώ δεν είναι μόνο θέμα ποινικού δικαίου, αλλά είναι και θέμα ε, πολιτικής μετανάστευσης και κοινωνικής πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν κοινό δρόμο, να εναρμονίσουν τις ε, νομοθετικές τους διατάξεις. Πρέπει να ενισχύσουμε την προστασία των θυμάτων, να μάθουμε η μία από την άλλη πλευρά για να ενισχύσουμε την πρόληψη. Εγώ λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα θα ακούσουμε την εμπειρία ε, πολλών οργανώσεων και πρωταγωνιστών σε αυτό το τομέα για να ε, καταλάβουμε ποια είναι η άποψή τους και τι πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού στην κοινωνία μας. Σας καλωσορίζω θερμά και εγώ από πλευράς μου. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να χαιρετήσω και μια ομάδα επισκεπτών ε, και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ ε, για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι χαίρουμε της ε, συνεχούς ε, υποστήριξη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ενισχύσουμε τον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων ε, και να συμπεριλάβουμε και νέα νομοθετικά μέτρα τόσο κατά την περίοδο πριν από την συνθήκη της Λισαβόνας και κατά την προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως και τώρα η ηθική αυτή υποστήριξη μπορεί να μεταφραστεί σε ένα χειροπιαστό ρόλο σε αυτήν την ε, διαδικασία ε, εκπόνησης ε, νομοθεσίας. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πλέον συνομοθέτης, νομοθετεί και αυτό εξίσου. Τα θέματα τα σημερινά είναι εντυπωσιακά, γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε θέματα νομικής και νομοθετικής φύσεως, παρότι βέβαια υπάρχουν και άλλοι τομείς ε, όπου αναπτύσσουμε πολλές δραστηριότητες. Όπως γνωρίζετε, η Κομισιόν η πρόταση της Κομισιόν που κατετέθη στα τέλη Μαρτίου για την ε, εκπόνηση οδηγίας νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εδώ πρόκειται για μια πρόταση που κατέγραψε στερή ιστορία γιατί κατατέθηκε μαζί με την οδηγία περί της ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Αυτό ήταν ένα πρώτο στοιχείο ε, ποινικού δικαίου που κατέθεσε η Κομισιόν μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και η κυρία Σοσίλια Μάλστρομ η Επιτροπός μας ε, θεώρησε ότι αυτή είναι μια σημαντική προτεραιότητα. Η πρόταση αυτή να είναι έτοιμη το συντομότερο δυνατόν. Και αυτό μάλιστα έγινε ένα μήνα μόλις μετά την ε, ανάληψη εξουσίας, ε, την ανάληψη του αξιώματος Επιτρόπου. Παράλληλα λοιπόν λάβαμε υπόψη μας τις συζητήσεις ε, που ε, λάμβαναν χώρα στο Συμβούλιο και προφανώς ε, το κείμενο έχει προσαρμοστεί στη συνθήκη της Λισαβόνας. Το κείμενο ακολουθεί ολιστική προσέγγιση, δίωξη των υπετίων, προστασία των θυμάτων. Αυτό βέβαια ήταν σαφές με βάση το ευρωπαϊκό ποινικό δικαίωμα και θέματα πρόληψης. Είμαστε λοιπόν ευγνώμονες στην Ισπανική Προεδρία για τον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τη συζητήση στο Συμβούλιο. Και αυτά ε, κατέληξαν, ε, οδήγησαν σε μια κοινή προσέγγιση την οποία υιοθέτησε το Συμβούλιο την ε, Παρασκευή της περασμένης εβδομάδας. Τώρα λοιπόν δρομολογείται η επόμενη φάση που προβλέπει ενδελεχή έλεγχο των κειμένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό χαιρετίζουμε αυτή τη συζήτηση που αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για ε, συζητήσεις. Συμμετέχουν ε, δύο επιτροπές, άρα δηλαδή είναι σαφές ότι θα αναπτυχθούν και δύο ε, διαφορετικές απόψεις, από διαφορετικό πρίσμα. Εμείς λοιπόν ως Επιτροπή είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε ότι το κείμενό μας δεν έχει αλλάξει ριζικά μετά από τις ε, συζητήσεις στο Συμβούλιο. Βέβαια, ελπίζουμε ότι οι συζητήσεις που θα γίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να επιφέρουν περαιτέρω βελτίωση. Τα θέματα που θίξαμε εμείς στο πλαίσιο των συζητήσεων Επιτρέψτε μου ε, ενδεικτικά να αναφέρω τρία θέματα. Το ένα είναι το θέμα της ε, της ετεροδικίας. Επίσης ε, το γεγονός ε, ότι οι δράστες ε, πολύ συχνά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολίτες μιας χώρας ε, και το έγκλημα γίνεται εκτός επικράτειας ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή το θέμα αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη νέα νομοθεσία. Δεν είναι δογματική προσέγγιση της Επιτρόπου που επιθυμεί διακαώς να συμπεριληφθούν παρέγκλητα κάποια στοιχεία της νομοθεσίας. Το θέμα είναι αποτελεσματική δίωξη και η δυνατότητα ανάληψης δράσης στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου. Βεβαίως, ε, προφανώς ε, προσφέρεται δωρεάν παροχή συμβουλών και αυτό πρέπει να επεκτείνεται σε όλα τα θύματα. Τέλος, αυτό που μπορεί να μοιάζει μια γραφειοκρατική και πληκτική λεπτομέρεια. Εμείς όμως θεωρούμε ότι αν τονίσουμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε περισσότερο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ε, για τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνουμε στοιχεία, με τον τρόπο αυτό θα είμαστε περισσότερο αξιόπιστοι. Και για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε ε, σωστή ενημέρωση από τα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι τα κράτη-μέλη ε, δεν επιθυμούν να επιβαρυνθούν ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα της ενημέρωσης, αλλά εμείς έχουμε την υποχρέωση να μεριμνήσουμε η ε, οδηγία να αποφέρει και αποτελέσματα. Ε, να πω και το εξής η Κομισιόν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα και ελπίζουμε ότι η συμφωνία ανάμεσα στα δύο νομοθετικά όργανα ε, η συμφωνία θα επιτευχθεί σύντομα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ομιλητές για σήμερα, γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να σταματήσω εδώ και να επιβεβαιώσω την ευγνωμοσύνη μας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σοβαρότητα με την οποία σε αυτή την υπόθεση. Ωραία. Πάμε τώρα στην Ισπανική ε, Προεδρία. Η Μαρτίνα Γκαρσία Ράντα έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Ε, θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι έρχομαι εκ μέρους του κυρίου Χωσέ Μολίνος και όχι εκ μέρους του κυρίου Λουίς Αγγέρα Ρουίς. Λοιπόν, εκπροσωπώ την Ισπανική Προεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συζητητές και την κυρία Μπάουερ για την οργάνωση του σεμιναρίου και την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω και την Επίτροπο Σεσίλια Μόρστρομ για την παρουσίαση της πρότασης ε, υπό τη δική μας Προεδρία, διότι αποτέλεσε ιδιαίτερη χαρά για μας να συνεργαστούμε και να χαιρετήσω και τις ε, ε, προσωπείς που στο πλαίσιο του Συμβουλίου κατέβαλαν προσπάθειες για να προωθηθεί αυτή η πρόταση και να οδηγηθούμε σε μια γενική συμφωνία στο Συμβούλιο Υπουργών ΔΕΗ στο Λουξεμβούργο την περσμένη εβδομάδα. Για να ξεκινήσω θα ήθελα να παρατηρήσω πως ε, αυτό του είδους τα εγκλήματα αφορούν και στην οδηγία του 2002 που αφορά την ευρωπαϊκή ρύθμιση σε αυτό το ζήτημα και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, περιέχει αυτό το οποίο περιείχε με η πρόταση του 2009 και που βασίζεται στα τρία π, δηλαδή στην πρόληψη, την δίωξη και την ε, ποινή, την κύρωση. Η πρόταση λοιπόν αυτή έχει ως στόχο την εναρμόνιση και προσέγγιση των εθνικών ε, νομοθεσιών και καθορίζοντας ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο μιλώντας για τις ε, μέγιστες ποινές και καταργήθηκαν ε, κάποιες άλλες ποινές οι οποίες την την προηγούμενη απόφαση πλαίσιο. Αυτό αποτελεί μια βελτίωση του νομοθετικού πλαίσιου και τεχνικής. Η προηγούμενη οδηγία αναφερόταν σε ποινές οι οποίες θα έπρεπε αναλογικές ε, και αποτρεπτικές. Η πρόταση τη οδηγία που παρουσίασε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Τροπή είχε ως στόχο την βελτίωση των δικαιωμάτων των θυμάτων παρέχοντας ε, μέτρα νομική αρρωγής αλλά και υποστήριξη. Μιλάω επίση και για ψυχολογική υποστήριξη, για ιατρική υποστήριξη αλλά και την ε, κατάρτιση, την εκπαίδευση των ανηλίκων ιδιαίτερα στα παιδιά των ε, θυμάτων. καθορίζονται λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα κάνει την, της ποινικής, ε, την ποινική διαδικασία και, τα, και ιδιαίτερα σε ό,τι φορά τα, τους ανήλικες θύματα βιασμών. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης και στην ρήτρα που αφορά την ευθύνη κάτι το οποίο αφορά στα οποία ή μάλλον να τονίσω ότι τα προληπτικά μέτρα αποτελούν μια καινοτομία. Περιέχεται η δυνατότητα χρήσης ε, των υπηρεσιών που ε, χορηγούνται στα θύματα σωματεμπορίας και εμπορίου λευκής σαρκός. Η ε, υλοποίηση ε, εκστρατιών ενημέρωσης και τέλος η κατάρτιση υπαλλήλων και των ατόμων τα οποία έχουν σε επαφή με τα θύματα. Τέλος, να τονίσω πως η πρόταση περιλαμβάνει κάποιες καινοτομίες όπως ε, το θέμα του ορισμού ε, των, της εμπορίας ανθρώπων, ε, την επέκταση της ετεροδικίας και καθορίζεται η υποχρεωτική ετεροδικία για τους υπηκόους των χωρών που διαπράττουν εγκλήματα εκτός των συνόρων και την χρήση κάποιων τεχνικών ανακριτικών και την νομιμοποίηση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αλλά και του ελέγχου των ε, κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών. Εμείς ε, αυτό που θέλαμε ήταν να πετύχουμε την συμφωνία στο Συμβούλιο, αυτό το κατορθώσαμε. Τώρα τα χέρια βρίσκονται στην ε, Κοινοβούλιο, αλλά και στην Βελική Προεδρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Βελγική Προεδρία τώρα. Σαλότ Γιάνσεν. Ευχαριστώ, καλή σας ημέρα. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και την Επιτροπή Γυναικών αλλά και τις εισηγήτριες κυρία Έντου και Μπάουερ για την πρόσκλησή τους και να μας κάτι που μας επιτρέψει να συμμετάσχουν στο το σεμινάριο για να σα αναφέρουμε τι προεδρίες, τη Πρωτεότητα τη Προεδρίας. Ε, το θέμα τη καταπολέμησης ε, τη ε, εμπορία ανθρώπου αποτελεί ένα βασικό στοιχείο του προγραμματό μα. Χαιρόμαστε που αυτή η οδηγία μπόρεσε να εγκριθεί από το Συμβούλιο ΔΕΗ την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτη προτεραιότητά μα, λοιπόν θα είναι να ξεκινήσουμε τον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φροντίζοντα ώστε ένας ανοιχτό και επικοδομητικό διάλογο, να μπορέσει να οικοδομηθεί και ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία ανάμεσα στα δύο όργανα ώστε το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων να ενισχυθεί το σύντομο δυνατόν. Από το δεκαετία του 1990 το Βέλγιο εργάζεται προκειμένου να καταπολεμήσει αυτό, αυτές οι εγκληματικές δραστηριότητες μια νομοθεσία η οποία προστατεύει τα θύματα και φυσικά ευθετήσαμε και μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που είναι θα έλεγα σφαιρική διότι περιέχει μέτρα πρόληψης, μέτρα προστασίας αλλά και μέτρα κατασταλτικά. Είναι ολοκληρωμένοι διότι έχουν δημιουργηθεί διάφορες δομές ώστε οι εμπλεκόμενοι και τα θύματα αυτών των και το υπεύθυνοι αυτών των ε, ζητημάτων να μπορούν να συναντώνται. Τώρα, η Βελγική Προεδρία θα οργανώσει ε, στις 18 και 19 Οκτωβρίου μια διάσκεψη. Τα θέματα της διασκέψεως ε, αφορούν ζητήματα επικαιρότητα και στηρίζονται επί των προτεραιοτήτων της προγράμματος της Στοκόλμης και το Action Oriented πρόγραμμα. Θα θέλαμε να δώσουμε λοιπόν με την ευκαιρία σε πολλούς εμπειρογνώμονες ε, γενικά λοιπόν η πρώτη μέρα του διασκέψεως ε, θα αφορά ζητήματα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας ε, τόσο σε εσωτερικό επίπεδο όσο και σε εξωτερικό και η δεύτερη μέρα θα αφιερωθεί σε ζητήματα που άπτονται της προστασίας των θυμάτων και στην πρόληψη. Πολλά ζητήματα θα εξεταστούν την δεύτερη μέρα. Μεταξύ αυτών το ζήτημα των κοινών προτύπων θα πρέπει να εφαρμοστούν σε ό,τι φορά την προστασία των θυμάτων αλλά και τις ιδιαιτερότητες για την προστασία των ανηλίκων. Το ζήτημα πρόληψης θα τονίσουμε ιδιαίτερα αφενός τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εκστρατιών ευαισθητοποίησης προκειμένου να υπάρξουν, υπάρξει καλύτερη στόχευση στις πρωτοβουλίες που χρειάζεται να ληφθούν στο μέλλον και στην ε, σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, το πρόγραμμα μας ε, σε ό,τι αφορά του επόμενου έξι μήνες ελπίζουμε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο και τον προβληματισμό πάνω σε ζητήματα καταπολέμησης ε, του ανθρώπινου εμπορίου. Uh, Καλά λοιπόν. Ε, εντάξει λοιπόν. Θα συνεχίσουμε στον επόμενο γύρο ομιλητών με εκπροσώπους της Ευρωπόλ, της Ευρωτζαστ και της Frontex. Παρακαλώ να ε, έλθουν να καθίσουν εδώ κοντά μας στο έδρανο του Προεδρείου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στον Στιβ Χάρβι που είναι εκπρόσωπος της Ευρωπόλ. Χάρβι κάπως μικρή καρέκλα μια στιγμή. Um, είναι, ωραίο αυτό το ανεπίσημο και συμπαθητικό περιβάλλον. Αλλιώς τα περίμενα. Πάντως αισθάνομαι να βρίσκομαι μεταξύ φίλων και πάντως συναδέλφων. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που απευθύνατε στην Ευρωπόλ για να προσέλθουμε εδώ δεν ξέρω πώς μου είχε ο κλήρος να μιλήσω πρώτος. Θα τα πω γρήγορα όμως. Η Ευρωπόλ είναι μια οργάνωση η οποία δεν δίνει τόσο το βάρος στην νομοθεσία. Εμείς υποστηρίζουμε τις δράσεις των χωρών μελών και μας δεσμεύει η εθνική νομοθεσία, οι χώρες μέλη επομένω. Και οι αποφάσεις και οι νομικοί μηχανισμοί που υπαγορεύουν το πώς δραστηριοποιούμαστε στην Ευρώπη. Είμαστε κυρίως οργάνωση η οποία παίζει ρόλο συντονιστικό συλλογή πληροφοριών και επιβολής του νόμου και της ε, τάξης. Ως οργάνωση και εγώ ειδικότερα ως εμπειρογνώμονας, όπως μου λένε κάποιοι άλλοι, για θέματα σωματεμπορίας, καλοδεχόμαστε κάθε πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον αγώνα κατά της σωματεμπορίας. Θα δώσω, θα ρίξω λίγο περισσότερο φως σε πιο παραδοσιακά στοιχεία. Για παράδειγμα, πώς να γίνει η, πώς γίνεται η παρα, παραδοσιακή αστυνόμευση. Για να τιμωρήσεις κάποιον πρέπει πρώτα να τον συλλάβεις, να τον πιάσεις. Άρα πρέπει πρώτα να συλληφθούν οι σώματέμποροι, να τους ασκηθεί δίωξη, να οδηγηθούν στα δικαστήρια πριν να καταλήξουν να τους επιβληθούν ποινές. Αν δεν τους συλλάβουμε, τους σώματεμπόρους, δεν θα πετύχουμε τον στόχο της προσπάθειάς μας να μειώσουμε δηλαδή τον τεράστιο αυτό τομέα παρανομία σε κάτι πιο εύκολα διαχειριστό. Οι σωματέμποροι είναι επαγγελματίες κακοποιοί. Προβαίνουν σε εκτίμηση των κινδύνων και αν δουν ότι οι κίνδυνοι είναι υπερβολική για αυτούς θα μεταθέσουν τις επιχειρήσεις τους αλλού. Όμως το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε για την ώρα δεν είναι εχθρικό για αυτούς. Διότι μπορούν και διαβαίνουν τα σύνορα των ευρωπαϊκών χωρών χωρίς μεγάλες δυσκολίες. Οι προσπάθειες των χωρών μελών έχουν βελτιωθεί βέβαια σημαντικά την τελευταία δεκαετία σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της σωματεμπορίας. Αλλά υπάρχει ακόμα χώρος για βελτίωση. Οι εθνικές ανταποκρίσεις, ας πω έτσι, είναι πολύ πιο έντονες από ό,τι παλαιά. Έχουμε έρευνες κατά των σωματεμπόρων σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει αυτό τώρα να περάσει στο επόμενο επίπεδο. Να υπάρξει περισσότερη διαμεθοριακή συνεργασία και διεθνείς έρευνες Αυτά θα συμβούν μόνον εάν υπάρξει συνειδητοποίηση ότι η έρευνα που γίνεται σε περιφερειακό, τοπικό, εθνικό επίπεδο μπορεί να περάσει σε ένα επίπεδο παραπάνω και μπορεί να γίνει επομένω και σε άλλη χώρα ή σε συνεργασία και με άλλη ή άλλες χώρες. Αυτό βέβαια από την πρώτη στιγμή δεν είναι πάντοτε προφανές. Από την ημέρα 1 ή εβδομάδα 1 εμείς η Ευρωπόλ θέλουμε να βλέπουμε οι πληροφορίες που συλλέγονται για τα δίκτυα σωματεμπορίας ή οι πληροφορίες που λαμβάνονται από όσους αναμειγνύονται σε αυτά ή από τα θύματα ή από άλλους εμπλεκόμενους. Θέλουμε αυτές οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις διάφορες αρχές να φτάνουν στην Ευρωπόλ αλλά και στην Interpol και στην Frontex και στη Eurojust στις οργανώσεις εκείνες δηλαδή που έχουν ιδρυθεί για να βελτιώσουν την διεξαγωγή των διαμεθοριακών ερευνών κατά του εγκλήματος, ώστε να μπορέσουν να ε, προχωρήσουν καλύτερα οι έρευνες αυτές. Αν λοιπόν τώρα θέλουμε, όπως είπα, να καταδικάσουμε τους σωματεμπόρους, πρέπει να συλλάβουμε και περισσότερους σωματεμπόρους. Ο τρόπος που θα το κάνουμε αυτό είναι διασφαλίζοντας ότι κάθε πληροφορία σχετική με τις δραστηριότητες αυτές να περνά στις υπεύθυνες ε, οργανώσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τις δραστηριότητε αυτές. Δεν πρόκειται για τίποτε μυστικές οργανώσεις. Ο ρόλος μας είναι δημόσιος. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι υπάρχει μια ε, σαφής έλλειψη συνειδητοποίησης στο χαμηλότερο επίπεδο. Δηλαδή, οι αστυνομικοί οι οποίοι ε, κάνουν τη δουλειά στα τοπικά και περιφερειακά και εθνικά επίπεδα δεν έχουν γνώση του ότι υπάρχουμε. Θέλουμε λοιπόν να βελτιωθεί η γνώση ότι υπάρχουν οι οργανώσεις αυτές στο ευρωπαϊκό επίπεδο που μπορούν να βελτιώσουν και τη δουλειά, να βοηθήσουν και τη δουλειά αυτού που εργάζεται στο τοπικό επίπεδο καθημερινά. Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα επιτρέψει την χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών για το σωματεμπόριο. Για πολλά χρόνια τώρα το σωματεμπόριο το χειριζόμαστε σαν κάποιο δίθεν μυστηριώδες έγκλημα. Οι ίδιες τεχνικές που, γίνονται, που χρησιμοποιούνται για την έρευνα για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, για το ναρκωτικό και για όλα τα σχετικά. Οι ίδιες χρησιμοποιούνται και εκεί, δηλαδή η, ε, η, η χρήση των παρακολουθήσεων τηλεφώνων, των πληροφοριοδοτών, των ε, αστυνομικών με πολιτικά και ούτω καθεξής. Τα ίδια πράγματα μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Δεν βλέπουμε όμως να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και διεξαγωγή ερευνών για το σωματεμπόριο και δεν γνωρίζω γιατί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν δίνεται προτεραιότητα στη σωματεμπορία όπως δίνεται σε άλλα εγκλήματα. Εάν δοθεί προτεραιότητα δεν θα επανερχόμασταν εμείς ξανά και ξανά σε βήματα όπως το δικό σας για να προσπαθήσουμε να προκαλέσουμε κάποια εντονότερη συνειδητοποίηση εάν υπήρχε η ίδια αντίδραση όπως για το εμπόριο ναρκωτικών. Βέβαια, κάνουμε πολύ περισσότερα σήμερα από ό,τι κάναμε ποτέ. Υπάρχουν όμως ακόμα πολλά βήματα που μπορούν να γίνουν. Όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου, η Ευρωπόλ είναι οργάνωση η οποία επιβάλλει τον νόμο και δεσμεύεται από την νομοθεσία και την εθνική, την ευρωπαϊκή και την διεθνή και τη δική μας νομοθεσία. Και δρούμε συμμορφούμενοι στην νομοθεσία αυτή. Ο ρόλο μα είναι να υποστηρίζουμε τι χώρε μέλη. Δεν έχουμε δύναμη καταναγκασμού, καμία εξουσία καταναγκασμού. Αυτά μπορούμε να κάνουμε, είναι προδιαγραμμένα από τον νόμο. Θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα και με την εμπλοκή των χωρών μελών, να μπορούν οι έρευνε και ανακρίσει μα να μπορέσουν να περάσουν και σε διαμεθοριακά. Ένα ε, μηχανισμό που χρησιμοποιείται ω παράδειγμα και χρησιμοποιείται περισσότερο τώρα, συχνότερα τώρα και είμαι σίγουρος ότι ο γείτονά μου θα μπορέσει να ε, συμπληρώσει και άλλα. Οι ομάδες ερευνητών που όλο και περισσότερες χώρες μέλη έρχονται στην Ευρωπόλη και στην Eurojust και υποβάλλουν ε, πρωτοβουλίες για την δημιουργία ομάδων, διεθνών ομάδων ε, προσώπων που θα διεξαγάγουν τις έρευνες με αποτέλεσμα να οδηγούνται στη δικαιοσύνη με πολύ αποτελεσματικότερο τρόπο. Δύο τέτοιες ομάδες που υποστηρίζει η Eurojust, μία για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρουμανία και ειδικά για την σωματεμπορία παιδιών, τα οποία ρίχνονται μετά στο έγκλημα στον δρόμο. Για ζητιανιά δηλαδή. Και χαίρομαι που τώρα αυτό έχει αναγνωριστεί ότι αποτελεί έγκλημα και αύριο θα ε, υπογράψουμε μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Βουλγαρίας σχετικά με Βουλγάρους υπηκόους οι οποίοι μεταφέρονται στον Ηνωμένο Βασίλειο για να ε, γίνουν πορτοφολάδες. Και αυτό έχει αναγνωριστεί πλέον ως έγκλημα και αυτό ε, ως έγκλημα δηλαδή που λαμβάνει μια ειδική προτεραιότητα και πάλι υπάρχει ομάδα στόχος που είναι τα παιδιά. Να λοιπόν δύο ομάδες που ε, θα αποδειχθούν πολύ σημαντικά εργαλεία για την ε, αντιμετώπιση διαμεθοριακά του εγκλήματος αυτού. Θα σας αφήσω με μια θετική νότα, κάνουμε πολύ περισσότερα, σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και με πολύ αποτελεσματικότερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Άρα τα νέα δεν είναι μόνο άσχημα, υπάρχουν και καλά νέα φτάνουμε σε ένα σημείο όπου γινόμαστε πλέον αποτελεσματικοί. Από τη δική μου σκοπιά πάντως ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε το εχθρικό περιβάλλον για τους σωματεμπόρους, για τους επαγγελματίες κακοποιούς, ώστε να τους αναγκάσουμε να σκεφτούν ξανά και ξανά πριν να προχωρήσουν στις παράνομες δραστηριότητες τους. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ε, διακόψουμε εντελώς το, ε, να, ε, σταματήσουμε εντελώς τη σωματεμπορία, αλλά μπορούμε να τους προκαλέσουμε δυσκολίες, να τους διακόψουμε τις ροές και ε, να τους ε, ε, αναχαιτήσουμε τον τρόπο αυτό. Ας μην μπω σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, προτιμώ να αρκεστώ σε αυτά και να είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις αν θέλετε αργότερα. Ευχαριστούμε κύριε Harvey. Στο τέλος ε, αυτών των εισηγήσεων θα ε, μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις. Τώρα έχει το λόγο η Όλα Λαουρέλ. Ο Όλα, με συγχωρείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτό το τόσο σημαντικό σεμινάριο. Εγώ είμαι ε, από τη Σουηδία αλλά ε, συμπτωματικά με Είμαι και ε, επικεφαλής της Eurojust ε, για τη σωματεμπορία και για την ε, προστασία των ανηλίκων. Εκπροσωπώ δηλαδή τη Eurojust ε, για θέματα προστασίας ανηλίκων. Πολύ σύντομα θα ήθελα να σας περιγράψω τα καθήκοντα της Eurojust. Φαντάζομαι περισσότεροι τα γνωρίζετε. Εμείς είμαστε η Ευρωπαϊκή Μονάδα δικαστικής συνεργασίας. Ε, συνεργαζόμαστε στενά με τη Europol και ο Στίβ έχει, σας ανέφερε, πολλά, πολλούς τομείς όπου αναπτύσσουμε κοινή δραστηριότητα. Εμείς ασχολούμεθα με σοβαρά εγκρήματα και εστιάζουμε στο οργανωμένο έγκλημα. Επίσης, δεν είμαστε απλά μια δικαστική οργάνωση για να υποστηρίζει θεωρητικά τη αντιμετώπιση του εγκλήματος. Το πράττουμε αυτό σε πρακτική βάση. Η συνεργασία ανάμεσα στις δικαστικές αρχές των κρατών μελών αλλά και τρίτων κρατών είναι σημαντικό εργαλείο για μας ένα σημαντικό εργαλείο για τη δίωξη στις χώρες όπου εμφανίζεται το έγκλημα. Εμείς λοιπόν ε, συνεργαζόμαστε και συντονίζουμε. Δηλαδή οι παλιοί μας ε, συναντιόνται στη Χάγη και αλλού για να μπορούν να συζητούν πώς θα αντιμετωπίσουν δύσκολες περιπτώσεις. Εξάλλου είμαστε κέντρο τεχνογνωσίας για τέτοιου είδους θέματα και οργανώνουμε και συναντήσεις που αφορούν θέματα βέλτιστης πρακτικής σε διάφορους ε, τομείς. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις ε, που αφορούν ε, στην εμπορία ανθρώπων, στα εγκλήματα κατά των παιδιών. Ίσως να έχετε δει τις πληροφορίες που είναι ανηρτημένες έξω από την αίθουσα. Και πρόσφατα δημοσιεύθηκαν και άλλες πληροφορίες. Μπορείτε να τις αποκτήσετε. Ας δούμε τώρα λιγάκι τις επιπτώσεις ε, της ε, νέας οδηγίας. Η Eurojust θα είναι σε καλύτερη θέση για να ε, μπορεί να διώκει την εμπορία ανθρώπων. Υπάρχουν πλέον και άλλες δυνατότητες. οι μέγιστες ποινές, αυτό είναι κάτι το καινούριο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι η νομολογία δεν ε, τοποθετείται μόνο στο θέμα της, ε, του εδάφους, της εντοπιότητας, αλλά και στο θέμα της προσωπικότητας. Θέλω να σας πω το εξής. Η Eurojust ε, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, όπου δηλαδή υπάρχουν ε, περιπτώσεις σύγκρουσης ε, δικαιοδοσίας, εμείς έχουμε τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους ε, τα προβλήματα. Ίσως να μοιάζουμε πολύ ήπιοι, αλλά εμείς όμως έχουμε το βλέμμα στραμμένο παρόλα αυτά στο οργανωμένο έγκλημα. Και γι' αυτό μας αφορά η δράση. Σε αυτήν θα εστιάσω την προσοχή μου στο υπόλοιπο της ομιλίας μου. Και θα αναφερθώ σε μία περίπτωση στη Γαλλία. Το 2004 οι γαλλικές αρχές ε, άρχισαν μία έρευνα μετά ένοπλη ληστεία που αναφέρθηκε στο νότο της Γαλλίας. Διακρύβωσαν λοιπόν ότι επρόκειτο για ε, ένα, μια ομάδα, οργανωμένη ομάδα εγκλήματος, που είχαν στη διάθεσή τους περίπου 100 γυναίκες που δούλευαν για αυτούς στην Ευρώπη. Η ένοπλη ληστεία ήταν εις βάρος τριών εκδιδόμενων γυναικών και η αστυνομία διαπίστωσε ότι υπήρχε κάποιος συσχετισμός, ε, κάποια σχέση ανάμεσα στη δουλειά των γυναικών και των επικεφαλής του οργανωμένου εγκλήματος που ήταν έγκλειστος σε φυλακή στη Βουλγαρία, όμως παρόλα αυτά μπορούσε από τη Βουλγαρία να κατευθύνει το δίκτυο μέσα από το κινητό του και ένα φαξ που είχε στη φυλακή. Ένας από τους ε, συγγενείς του ήταν επίσης στην κεφαλή της ομάδας και μία από τις γυναίκες η οποία ήταν θύμα κατά τη διάρκεια της ένοπλης ε, ληστείας και αυτή ήταν μέλος της οργάνωσης. Η όλη λοιπόν ιδέα ήταν η εξής. Μία γυναίκα να έχει στη διάθεσή της ένα κελί και ένας άνδρας να διαθέτει μια σειρά τέτοιων ε, μονάδων που εντοπίστηκαν ε, στην Αυστρία, στην Ισπανία, στην Ολλανδία μεταξύ άλλων. Αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα ε, βίαιες μεθόδους για να έχουν υπό τον έλεγχό τους τις γυναίκες. Απαγωγή, απειλές, βία, ακόμα και ε, ανθρωποκτονίες. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες τις μετακινούσαν ε, στις διάφορες πόλεις και οι γυναίκες αυτές δεν παρέμεναν σε μια πόλη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά από λίγο καιρό μετακινούνται αλλού. Και υπάρχει ένα παράδειγμα. Μία ε, εκδιδόμενη γυναίκα άρχισε να δουλεύει στην ηλικία των 18 ετών ε, και πριν διαλυθεί το δίκτυο είχε δουλέψει στο Μιλάνο, στο Μονπεγέ, στη Λιόνι, στο Ρότερνταμ, πάλι στη Λιόν και μετά στο Μονπελιέ. Το 2007 οργανώστηκε συντονισμένη επίθεση μεταξύ ε, Γαλλίας, Ιταλίας και Βουλγαρίας. Και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ε, παρατήρηση σε αυτή την περίπτωση. Αυτές οι γυναίκες δούλευαν στο χώρο της ε, νόμιμης πορνείας. Πολύ συχνά βέβαια αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει ο πελάτης αν δεν το ρωτήσει. Και ο πελάτης δεν ρωτάει γιατί δεν θέλει να ξέρει. Δεν ξέρει αν είναι έγκλημα. Ε, γιατί αν είναι έγκλημα η εκδιδόμενη γυναίκα προφανώς κανείς δεν θα ρωτήσει και δεν θα ήθελε να βρεθεί κάποιος στο δικαστήριο που να μπορεί να το αποδείξει αυτό η εκδιδόμενη. Οι γυναίκες αυτές δεν επέλεξαν ε, το επάγγελμα που ασκούν. Στην περίπτωση αυτή οι γυναίκες εξαναγκάστηκαν στην πορνεία. Πολύ λυπηρό αυτό, αλλά δυστυχώς ε, σήμερα στην Ευρώπη ε, συχνά οι, προστι... οι εκδιδόμενες γυναίκες είναι σε ομοιρία, ε, σε, σε κατάσταση σωματεμπορίας. Όλα αυτά έγιναν το 2007. Η Γαλλία εξέδωσε 13 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης που είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο. Από το 2002 έως το 2006 αυτή η εγκληματική οργάνωση ε, προσπορίστηκε 10 εκατομμύρια ευρώ. Οι γυναίκες ε, μπορούσαν να κρατήσουν το 30% αν ήταν παραγωγικές ε, και υποταγμένες. 70 έπαιρνε η οργάνωση και το 20% το κρατούσε ο επικεφαλής. Ε, χρησιμοποίησαν τη Western Union για να μεταφέρουν τα χρήματα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν από την Western Union. Χρησιμοποίησαν επίσης ε, δομές επιχειρηματικές στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες για να ξεπλύνουν το χρήμα. Έτσι λοιπόν ε, το μαύρο χρήμα τελικά με το ξέπλυμα έγινε άσπρο. Η Γαλλία εξέδωσε εντάλματα, ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης ε, κατά δύο από την ομάδα. Αυτή βέβαια εξέτειαν ποινή για το ίδιο έγκλημα στη Βουλγαρία. Και η Βουλγαρία ισχυρίστηκε ότι δεν είναι δυνατόν να διωχθούν διότι η πρώτη καταδίκη καλύπτει και τη δεύτερη, το, τη γαλλική, νέμπι να Έτσι λοιπόν η νεπλάκη Eurojust και η Γαλλία ε, ζήτησε από τη Eurojust ε, αρρωγή. Έλαβαν χώρα πάρα πολλέ επαφέ, άτυπε και επίσημε ανάμεσα στους συνεργάτες μας. Η Eurojust οργάνωσε μία συνάντηση συντονιστική που όπως σας είπα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Έτσι λοιπόν οι ε, ανακριτές και οι δικαστές ε, είχαν πλέον την ευκαιρία να συζητήσουν. Αποτέλεσμα. Η Γαλλία κατόρθωσε κατά τη διάρκεια της συνάντησης να αποδείξει ότι τα εγκλήματα στη Γαλλία δεν καλύπτονται από την καταδίκη στη Βουλγαρία και τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης τα οποία εστάλησαν στη Βουλγαρία έγιναν αποδεκτά. Με αποτέλεσμα το 2008 οι δύο βασικοί ύποπτοι να εκδοθούν στη Γαλλία ε, προσωρινή έστω έκδοση κατά τη διάρκεια της έκτησης της ποινής. Το 2008 είχαμε τις συνεντεύξεις ε, στη φυλακή στη Γαλλία και το 2009 ε, καταδικάστηκαν σε 8 και 9 χρόνια αντίστοιχα. Τώρα το 2010 επανήλθαν στην Βουλγαρία για να εκτίσουν το υπόλοιπο της ποινή τους στη χώρα αυτή. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα για το πώς ε, δουλεύει πρακτικά η Eurojust και έχω και κάποιες ε, πληροφορίες που αφορούν σε επαφές αυτής της ε, και στο σημείο επαφή που μπορεί κανεί να απευθυνθεί για την προστασία των παιδιών. Υπάρχει και μια ιστοσελίδα που δείχνει τη δουλειά τη Eurojust σχετικά με την προστασία των παιδιών και μπορεί κανεί ε, να προσφύγει σε αυτήν μέσα ε, με link από την ιστοσελίδα τη Eurojust. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λόρελ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Άννα Κριστίνα Χόρχε από την Frontex. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Άννα Κριστίνα Χόρχε, έρχομαι από την Frontex ε, στις Βρυξέλλες, ε, είμαι εξωματικός σύνδεσμος. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή και τους εισηγητές που με επέτρεψαν να συμμετάσχω σε αυτό το σεμινάριο και να μου δίνετε ευκαιρία να σας μιλήσω. Τώρα το θέμα της σωματεμπορίας ε, δεν είναι ένα θέμα που αφορά την Frontex ε, άμεσα σύμφωνα με την ε, απόφαση του 2005-2007. Έχουμε εμεί στόχο να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση μέσω συνεργασία των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα της Frontex. Η Frontex λοιπόν ε, οργανώνει τη δραστηριότητά της σε ό,τι φορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ε, συνεργασία για να μειώσει αυτό το φαινόμενο. Πάντως, ότι η σωματεμπορία θεωρείται ότι αποτελεί ένα σοβαρό οργανωμένο έγκλημα και βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της ε, Europol αναγνωρίζουμε ότι τα σήματα αυτού του είδους των δραστηριοτήτων, δια, διασχίζουν τα σύνορα, βοηθούμενοι από τους ε, σωματεμπόρους και αναγκάζουν τις ε, διάφορες οργανώσεις να αντιδράσουν σε αυτή την δραστηριότητα. Αυτό ε, αναγνωρίστηκε μάλλον κατά διάρκεια διαφόρων δραστηριοτήτων για την προστασία θυμάτων σωματεμπορίας. Επίσης, σαφές αποτέλεσμα από τις ε, εργασίες της Frontex ε, μετά από την πίεση που ε, επήλθε στα σύνορα. Η διάφορες δραστηριότητε ε, που πρόθεσαν οι προεδρίες ε, του Συμβουλίου σε διάφορες μορφές και σε διάφορους μορφότυπους συνδέεται με δραστηριότητε ε, για την αξιολόγηση και κατανόηση του φαινομένου από τα κράτη-μέλη του 2006 η Προεδρία της Αυστρίας επικεντρώθηκε στην σωματεμπορία και ε, πρόθεσε την ε, αναζήτηση διακριμένων στοιχείων. Η συνεργασία με την Europol και την Interpol συνέβαλε στην δημιουργία δικτών συγκρίσιμους μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων και πρωτοβουλειών ήταν διαδικασία κατάρτισης που πρόθεσε η Σουηδική Προεδρία, η οποία οδήγησε παράλληλα με το πρόγραμμα της Στοχόλμης να καταρτιστεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας. Κατά διάρκεια λοιπόν αυτού του σχεδίου, η Europol, Eurojust και η Frontex ε, προσπάθησαν να βελτιώσουν τη συνεργασία του για την καταπολέμηση. Το έγγραφο αυτό χρησιμοποιεί μια σαφή γλώσσα για την ανάγκη περαιτέρω συνεργασία ε, των οργάνων σε αυτόν τον τομέα πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, στο οποίο συμμετέχει και η Frontex ε, μέσω διάφορων πιλωτικών σχεδίων. Η Ισπανική Προεδρία αποφάσισε να ε, διατηρήσει την στόχευση σε αυτό το θέμα και ε, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τους ασυνόδους ανηλίκους του πιο ευάλωτος ε, στο ζήτημα της εμπορίας. Ζητήθηκε από την Frontex να κάνει ανάλυση, συλλογή στοιχείων αλλά και να ανάλαβει δραστηριότητε στον τομέα. Όλα αυτά λοιπόν είναι δραστηριότητε κλειδί για τις μελλοντικέ δραστηριότητε σε αυτόν τον τομέα η Επιτροπή για την Εσωτερική Συνεργασία, ΚΟΖΗ, όπως και το Συμβούλιο, είναι, συζήτησαν ήδη συστάσεις σχετικά με την έκθεση της Μαδρίτης, που, στοχεύεται, που βασίζεται συγγνώμη, στην, στο αποτέλεσμα της Europol και στην ε, αξιολόγηση κινδύνου προκειμένου να προληφθεί η σώματεμπορία στα εξωτερικά σύνορα της κοινότητας. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, η επικείμενη Βελική Προεδρία θα συνεχίσει να βασίζεται στο κείμενο της Στοχόλμης και προσβλέπει στην διάσκεψη η οποία θα γίνει όπως γνωρίζετε τον Οκτώβριο του 2010. Το Frontex υποστηρίζει και τη Βελική Προεδρία και το κέντρο για την Ευρωπαϊκή Διεθνή Δράση μετά την προετοιμασία και διοργάνωση αυτού του σημαντικού γεγονότος το οποίο θα ασχοληθεί με το ζήτημα της ε, σωμπατεπορίας και της ε, επιβολής του νόμου. Η Frontex λοιπόν αυτό το οποίο φροντίζει είναι να εφαρμόσει όλα αυτά τα προγράμματα με τον καλύτερο τρόπο. Η Frontex λοιπόν έχει αναπτύξει και ένα πιλωτικό σχέδιο που περιλαμβάνει τις, ε, τα βασικά στοιχεία που αφορά την ε, συλλογή στοιχείων το 2008 από κοινού με τα κράτη-μέλη και τη συμμετοχή της Europol και άλλων διεθνών οργανώσεων δημιουργήθηκαν κάποιοι δείκτες ε, αυτό το αρχικό σχέδιο λοιπόν συνεχίστηκε το 2009 και οδήγησε στα παρακάτω αποτελέσματα. Ε, δείκτες ε, ετήσιους για την συλλογή στοιχείων, μια συλλογή στοιχείων για τις κοινέ ε, δράσεις, ε, την ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί και μια επιπλέον ανταλλαγή ε, στοιχείων με την Europol και με άλλες διεθνείς οργανώσεις. Το βασικό όμως είναι ότι δημιουργήσαμε και ένα προφίλ ε, των ε, διακινητών. Αυτό βασίζεται σε συλλογή στοιχείων από τα 27 κράτη-μέλη και καλύπτει το έτος 2008. Μας δίνει μια γενικότερη άποψη για την σωματιμπορία στην στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων ε, υπογραμμίζει τις ε, βασικές εθνικότητες που κινδυνεύουν να καταστούν τα σώματα εμπορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνει σε ποιες ε, χώρες γίνεται μεγαλύτερη διακίνηση και που έχουν εντοπιστεί οι διακινητές. Επίση, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει δυσκολίε σε ό,τι αφορά του συγκρίσιμου ορισμού σε εθνικό επίπεδο, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε διπλή ε, καταμέτρηση και κάτι το οποίο στρεβλώνει την εικόνα. Πάντως αυτή η εικόνα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις αρχές συμβουλής της τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι καθορίζει τα προφίλ των διακινητών. Αυτά τα προφίλ αποτελούν την βάση για την βελτίωση της ευαισθησίας και την πρόκληση κάποιων πληροφοριών σε σημαντικού ε, συνδέσμους διότι ε, αυτοί είναι οι πρώτοι από όλους που μπορούν να βοηθήσουν ε, τα θύματα. Τώρα, σε άλλους τομείς η Frontex αναπτύσσει διάφορες θεότητες κατάρτισης, διότι σύμφωνα με την νέα πρόταση οδηγίας για την πρόληψη και κατεπολέμηση της οματεμπορίας και την προστασία των θυμάτων αυτής, τα κρατημέλη θα πρέπει να προάγουν μια ε, κατάρτιση των ε, αξιωματικών για την προστασία των θυμάτων συμπεριλαμβανομένων και των ε, συνοριοφυλάκων και η Frontex με την μισθανθία της ΥΠΟΛ προσπαθεί να εφαρμόσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις προτάσεις. Και να πω τώρα κάτι για την Frontex ακόμα, για μια πρόταση που είχε κάνει η Κομισιόν τον Φεβρουάριο 2010, την αναθεώρηση του κανονισμού Frontex. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά την άδεια πραγμάτευση, η οποία θα λάβει χώρα και στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο και να τονίσω ότι Όπως όλοι γνωρίζετε, η Frontex ε, δεν είναι σε θέση να επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία. Πάντως, ε, και αυτό το είπε και ο συνάδελφος από την Europol, ε, δηλαδή τη σημασία που έχει η ανταλλαγή προφοριών, ειδικά στον τομέα της ζώματεμπορίας όταν εντοπίζουμε ενδυνάμει διακινητές στα εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, μεταξύ Europol και Eurojust αλλά και μεταξύ των εθνικών ε, αρχών επιβολής του νόμου. Συζητώντας λοιπόν αυτό το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, θα ήθελα να λάβετε υπόψη ότι η Frontex ε, χρειάζεται αυτά τα στοιχεία για δικούς τους λόγους, πρώτα για να κάνει την ανάλυση κινδύνου και ως εκ τούτου να μπορέσει να οργανώσει και να αναλάβει ε, εστιασμένες δράσεις, αλλά αυτά τα στοιχεία φυσικά δεν τα επιθυμούμε μπορούμε να τα καταχωρήσουμε και να τα αποθηκεύσουμε σε κάποιες βάσεις δεδομένων. Θέλουμε να ενισχύσουμε λοιπόν τις δυνατότητες που έχουμε για τη συλλογή στοιχείων σε περιπτώσεις ε, ερευνών, ε, ανακρίσεων και δίωξης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας και, και οι τρεις παρεμβάσεις. Θα δώσω τον λόγο τώρα για την διεξαγωγή συζητήσεως στα πρόσωπα που βρίσκονται στην αίθουσα. Παρακαλώ όμως όλες και όλους να περιοριστούν σε δύο λεπτά εάν θέλουν να κάνουν κάποια ερώτηση. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην Αναγκόμες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για αυτή την πρωτοβουλία του να ε, συνεργαστεί εδώ η Επιτροπή με τους ε, Και θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον από τους τρεις ε, ομιλητές μήπως γνωρίζουν κατά πόσον υπάρχει μία ομάδα που να είναι ιδιαίτερα τρωτή ε, αναφέρομαι στα μωρά τα οποία απάγονται μέσα από συγκαλυμμένες ε, απαγωγές δίθεν ε, πλασματικής υιοθεσίας. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ε, Ρουμανία, νομίζω και την Ουγγαρία. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω κατά πόσον έχετε να μας πείτε κάτι για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε να κάνουμε με ε, οργανωμένο έγκλημα, ομάδες οργανωμένου εγκλήματος ε, που ε, αναζητούν τρόπους συγκαλυμμένους για να αποφύγουν τη δίωξη, όπως συμβαίνει με τη σωματοπορία. Και μήπως ξέρετε κάτι γι' αυτό που ρώτησα εγώ. Επίσης, μήπως γνωρίζετε κάτι το κατά πόσο είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί στην οδηγία το θέμα της ετεροδικίας. Κοιτάξτε, γνωρίζουμε περιπτώσεις όπου Ευρωπαίοι ε, ενεπλάκησαν στην ε, εμπορία παιδιών από άλλες χώρες. Μία περίπτωση πρόσφατα αυτή που δεν ήταν ε, ευρωπαϊκή αλλά αμερικανική και είχαμε μια άλλη περίπτωση στο Τσάντ πριν από περισσότερο καιρό για παιδιά που απήχθησαν αλλά δεν ήταν ορφανά αυτά τα παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι ε, ε, διώχθησαν επειδή ε, συμμετείχαν σε αυτό το κύκλωμα. Τι έχετε να μας πείτε από αυτού. θα ήθελα καλύτερα να συγκεντρώσουμε ερωτήσεις και μετά στο τέλος να απαντήσουν οι ομιλητές. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Σίλβια Κώστα και παρακαλώ να έχετε κατά νου ότι για δύο λεπτά μπορείτε να μιλήσετε για να μπορέσουν να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Ε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτά που μας είπατε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τρεις ερωτήσεις πολύ σύντομες. Η πρώτη είναι η εξής. Εσείς ε, το πρώτο βήμα για να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία που είναι πολύ σημαντική δεν πιστεύετε ότι το πρώτο σημαντικότερο είναι να εναρμονίσουμε το πλαίσιο του 2004 που αφορά στην άδεια παραμονής και που ήταν συνάρτηση με το κατά πόσο είναι κανείς θύμα ή όχι. Γιατί η εμπειρία ε, μας δείχνει ότι ακόμα και αν υπάρχει καταγγελία για μία βίαιη πράξη θα πρέπει να υπάρχει και αρρωγή. Κοιτάξτε, Στη δική μου τη χώρα και άλλοι θεωρούμε ότι πρέπει οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να συνεργαστούν με της ΜΚΟ, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ε, υποδοχή και στην ε, συνεργασία με τις ε, δυνάμεις ασφαλείας της ένωμης τάξης και βοήθησαν στην επαναπρόθεση. Τελευταία ερώτηση. Εσείς μιλήσατε για σημαντικά εργαλεία και θέλω να πω το εξής. Στη δική μου τη χώρα, δυστυχώς, πάμε προς τα πίσω όσον αφορά τις υποκλοπές και αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο κατά τη γνώμη μου. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό. Εδώ δεν γίνεται και λόγος για το ε, έγκλημα στον κυβερνοχώρο, κυβερνοέγκλημα που παίζει ρόλο στη σωματεμπερία και παίζει, χρησιμοποιεί και το διαδίκτυο. Ίσως να υπάρχει κάποιο άλλο εργαλείο. Αλλά από αυτά που μας είπατε νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα ε, το οποίο θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη στην κατάρτιση της οδηγίας. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό? Η κυρία Κορνέλια Ernst. Δύο πράγματα. Πρώτα θέλω να ρωτήσω την κυρία της Frontex Πρέπει να γίνει σαφή διάκριση ανάμεσα σε σώματεμπορία, δηλαδή εμπόριο φυσικών προσώπων. Και ε, μέσα στο σχέδιο υπάρχει ένα άρθρο 2, όπου λέει, αναφέρεται πραγματικά, για ε, σκοπούς εγκληματικότητας και με χρήση βίας και απάτης κτλ. Μιλάμε δηλαδή για ανθρώπινες δράσεις. Αυτό είναι άλλο όμως από την παράνομη μετανάστευση Είπατε ότι ισοδυναμεί με παράνομη μετανάστευση. Είναι το ίδιο για εσά. Άλλο το λαθρεμπόριο ανθρώπων και άλλο η σωματεμπορία. Πώς τα χειρίζεστε αυτά κάνοντας μια διάκριση ανάμεσά τους. Δεύτερο, η ζητιανιά όταν βγαίνουν τα παιδιά στους δρόμους να ζητιανεύσουν. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό γιατί και σωστά, και σωστά μπαίνει εδώ ως εκμετάλλευση, δεν υπάρχει θέμα, αλλά πώς ε, γίνεται η δίωξη, πώς ε, γίνεται η έρευνα, για μένα είναι πολύ προβληματικό. Η κυρία Τόμσεν, ευχαριστώ, ευχαριστώ και για τις παρουσιάσεις σας. Να ρίξουμε μια ματιά και στην πλευρά της ζήτηση των υπηρεσιών. Είπα ότι θα γίνει ένα είδος ταξινόμησης. Τι είδους υπηρεσίες πρόκειται να ποινικοποιηθούν. Και ο κύριος Λαουρέλ, για σας είναι η ερώτηση Είπατε ότι είναι δύσκολο να ποινικοποιηθούν οι πελάτες, γιατί οι ίδιοι οι πελάτες δεν ρωτούν την ε, ε, πόρνη εάν είναι νόμιμη παράνομη. Ούτως ή άλλως όμως αυτό δεν πρόκειται να τους αποτρέψει από του να ε, χρησιμοποιήσουν τι υπηρεσίε τη γυναίκα, γιατί έχουμε δει στη Δανία την πατρίδα μου πολλές περιπτώσεις όπου ο πελάτης του το λέει η ίδια γυναίκα και λέει καλά δεν με ενδιαφέρει εμένα και εκεί ε, η πορνεία έχει γίνει ολόκληρη, ολόκληρη βιομηχανία. Δεν είναι αποτρεπτικό λοιπόν, αντίθετα μάλιστα. Πώς νομίζετε λοιπόν ότι μπορεί να θεσπιστεί κάποια νομοθεσία η οποία να ποινικοποιεί την ιδιότητα του πελάτη Άλλωστε η κατάσταση αυτή συναντάται και στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χώρων. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες με τις οποίες ε, βοηθάτε και εμάς σήμερα να έχουμε έτσι μια γενικότερη εικόνα σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτού του τόσο σοβαρού προβλήματος. Ε, δημοσιεύτηκε σήμερα μάλιστα μια παγκόσμια έκθεση από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών στην οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 155 χώρες. Και η ερώτησή μου είναι λίγο πιο ευρεία σε σχέση με τον συναδέλφων ε, αναφορικά με ένα μέγεθος που έχει αυτή η έκθεση. Αναφέρεται λοιπόν ότι καταδικαστικές αποφάσεις στις περισσότερες από αυτές τις χώρες ε, δεν υπερβαίνουν ανά 100.000 άτομα έχουμε μόνο μια μισή απόφαση. Σε 100.000 άτομα έχουμε μόνο μια μισή απόφαση. Και διαρωτώ με, ενώ εντείνουμε την προσπάθεια, ενώ φαίνεται ότι δημιουργούμε επιπρόσθετους μηχανισμούς, το πρόβλημα τελικά αναφέρεται στις δομές μας, αναφέρεται στις διαθροτικές δομές σε κάθε κράτος μέλος και ευρωπαϊκά ή πρέπει να δώσουμε έμφαση και στην πολιτική βούληση που πρέπει να υπάρχει στο μέλλον. Μήπως υστερούμε στην πολιτική βούληση και εμείς όλοι οι συνάδελφοι και τα κοινοβούλια τα εθνικά πρέπει να τονίσουμε αυτή την πτυχή του προβλήματος. Σας ευχαριστώ. Uh, Το εμπόριο ανθρώπων είναι κάτι πολύ διαφορετικό από οποιαδήποτε ε, κανονική ε, οικονομική δραστηριότητα αφού καθιστά τα πρόσωπα αντικείμενα ή οικονομικούς πόρους αν θέλετε. Όντως ο σύγχρονος καπιταλισμός ε, προσλαμβάνει και απολύει πρόσωπα ανθρώπους όπως θέλει, όπως κάνει άλλωστε και ο σωματέμπορος. Η παράνομη σωματεμπορία, η ε, πρόσληψη σε υπεράκτες, ε, μέσω υπεράκτων εταιριών και ούτω Όλα αυτά είναι φαινόμενα, όλα αυτά είναι πλευρές του ίδιου φαινομένου. Και η σωματεμπορία ανθεί σε ένα κλίμα όπου οι άνθρωποι θεωρούνται ως οικονομικοί πόροι. Αυτό το κλίμα πρέπει να αλλάξει πρώτα-πρώτα. Αποκαλυπτικό ήταν το ότι η κυρία της Frontex νομίζω είπε ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες από τις οποίες προέρχονται τα περισσότερα θύματα και υποθέτω βέβαια ότι θα είναι χώρες με πολύ χαμηλό εισόδημα ή ε, ε, επίπεδα αμοιβών. Διαρωτώ με εάν ε, τα, τα θύματα προέρχονται κυρίως από ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να το μάθει κανείς. Αποκαλυπτικό επίσης μου φάνηκε ότι φαίνεται πως η συμφωνία Σέγγεν και κυρίως η κατάργηση των συνόρων έχει διευκολύνει την σωματεμπορία. κυρία Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Ευχαριστώ για τις ε, παρουσιάσεις σας. Βέβαια, είναι πολλές ερωτήσεις που έχω αλλά θα περιοριστώ σε τρεις και σύντομες. Ποιοι είναι οι παρόντες υπολογισμοί του όγκου του σωματεμπορίου στην Ευρώπη. Επίσης, ποιες είναι οι νέες τάσεις, εάν υπάρχουν, εάν σημειώνονται νέες τάσεις στη σωματεμπορία. Την τελευταία φορά δηλαδή που είχαμε ασχοληθεί με το θέμα, η τάση που διαμορφωνόταν ήταν ότι κυρίως το λαθρεμπόριο ανθρώπων για την αγορά εργασία ήταν αυτό που είχε περισσότερη ε, ζήτηση ας πούμε. Ποια είναι σήμερα η κατάσταση. Και η τρίτη μου ερώτηση αφορά την διακίνηση προσώπων μέσα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, για τι αριθμούς μιλούμε και ποιες είναι οι οδοί ή και ποια είναι τα είδη της ε, εμπορίας ανθρώπινων όντων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κάπου έχω την αίσθηση ότι όλες μας οι προσπάθειες κατευθύνονται στην καταπολέμηση των ροών αυτών που προέρχονται από τρίτες χώρες και ίσως ρίχνουμε, λιγότερη, προσοχή στο τι συμβαίνει μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένω τις απαντήσεις σας. Τελευταία ερώτηση. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τις σημαντικές σας παρουσιάσεις και ως εισηγήτριας από πλευρά Επιτροπή των Γυναικών για την ε, προστασία θυμάτων πρόκειται για μια έκθεση την οποία καταρτίζουμε θεωρώντα ότι τα θύματα θα πρέπει να προστατεύονται με τον αυτό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και πέραν του ότι τα άτομα θύματα σωματεμπορίας, ε, ανθρώπινη εμπορία ε, προστατεύονται από μια οδηγία θα ήθελα να σα κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Εγώ στο εκτιμώντας Έχω συμπεριλάβει κάποια στοιχεία που αφορούν στα θύματα και η ερώτησή μου λοιπόν έχει ως εξής. Πιστεύετε ότι όντως μπορούν να προστατευτούν μέσω αυτής της οδηγίας και κατά πόσο θα ήταν χρήσιμο από τη στιγμή που θα πρέπει να υπάρχει κάποιος γνωστός διακινητής και μιλώντας για οργανωμένο έγκλημα, έχουμε κάποιον άτομο το οποίο γνωρίζουμε την ταυτότητα. Ευχαριστώ. Tack ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές για να απαντήσουν ε, θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη συγκέντρωση ε, δεδομένων πρώτα απ' όλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και μετά σε διεθνές επίπεδο. Γιατί αν θέλουμε να προχωρήσουμε ε, πρέπει καταρχήν να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του πώς ε, λειτουργούν τα πράγματα στα κράτη-μέλη. Και εδώ θα ήθελα να πω το εξή σχετικά με τη Frontex. Είπατε ότι πρέπει να εκπαιδευτούν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο μέλλον. Ελπίζω λοιπόν ότι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης αυτής μπορούμε και να αποκτήσουμε μια εκπαίδευση εστιασμένη στα παιδιά και τις γυναίκες. Γιατί κατά κύριο λόγο αυτοί είναι τα θύματα της σωματεμπορίας. Θα τώρα να δώσω το λόγο ε, στους ομιλητές για να απαντήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάω με την τελευταία ερώτηση. Η Europol είναι σε θέση να συγκεντρώνει δεδομένα και τα κράτη-μέλη ε, γι' αυτό τον λόγο καταφεύγουν στη Europol. Εχθές, παραδείγματο χάρη, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση. Ο Στίβ ίσως ε, μπορεί να ε, τοποθετηθεί σε αυτή την περίπτωση. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε νέες αποφάσεις και εκείνο που ενδιαφέρει είναι να συγκεντρώσουμε δεδομένα από τα κράτη-μέλη που θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν, ε, θα μας προσφέρουν ε, στο μέλλον ε, ένα καλύτερο όπλο, αποτελεσματικότερο όπλο για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τις υιοθεσίε, εξ όσων γνωρίζω, αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Η υιοθεσία ως μέσον σωματεμπορίας, αυτό δεν είμαστε αρμόδιοι εμείς γι' αυτό. Ως προς την απλούστευση των πραγμάτων ε, υπάρχουν πάρα πολλές ε, δυνατότητες ε, μπορούμε να δούμε λιγάκι του τους σωματέμπορους, τους λαθρέμπορους οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα κενά στις νομοθεσίες των κρατών μελών για να εντοπίσουν παραθυράκια. κατόπιν, ετέθη μία ερώτηση σε μένα, κατά κύριο λόγο σε μένα, σχετικά με τη ζήτηση. Εγώ θέλησα να πω το εξής, ότι αν ποινικοποιήσουμε τον πελάτη που αγοράζει σεξ, σεξουαλικές υπηρεσίε από το θύμα σώματεμπορίας και μπορεί κανείς να το αποδείξει, τότε η νομοθεσία πάβει να έχει σχή πολλοί στην αρχή ήταν υπερήφανοι που έχουν αυτή την νομοθεσία. Αν όμως ε, ερωτήσει κανείς σε τελική ανάλυση πόσοι διώχθηκαν, πόσοι καταδικάστηκαν, δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός. Εγώ λοιπόν δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όταν μιλάμε για ε, νόμιμη πορνεία, αυτό μπορεί να σας μοιάζει κάτι το αποδεκτό, αλλά μην ξεχνάτε ότι το 80% των γυναικών που εργάζονται σε αυτό το χώρο της νόμιμης ε, πορνείας ε, οι περισσότερες εξ αυτών είναι θύματα σωματεμπορίας. Εγώ λοιπόν πιστεύω το εξής και αυτό το λέω σε εκπρόσωπος της Eurojust. Εγώ θεωρώ ότι το να ποινικοποιηθεί η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, δεν γνωρίζω τίποτα από αυτόν. Ε, ενδιαφέροντα ηχούν. Όταν ε, προβαίνει κανείς στην εναρμόνιση, η εναρμόνιση ε, είναι πολύ πιο αποτελεσματική εάν παρέμενε κανείς ε, απλά αρμόδιος σε ένα και μόνο κράτος μέλος. Λοιπόν, ελπίζω να κατέγραψα όλες τις ε, ε, ερωτήσεις με τη σειρά που Όσον αφορά τα μωρά, υπάρχουν πολλές έρευνες που αφορούν την σωματεμπορία γυναικών στο τελικό στάδιο της εγκυμοσύνης για να εκμεταλλευτούν αργότερα και τα μωρά. Αυτό δεν είναι ο κύριος όγκος της σωματεμπορίας, αλλά υπάρχει και αυτό και μερικοί εστιάζουν εκεί την προσοχή τους. Ε, γιατί αποδίδει αυτή η ενέργεια. Έχουμε απογοτευμένους ε, υποψήφιου εν δυνάμει γονεί που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν πολλά χρήματα για να αποκτήσουν παιδί. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω, οι σωματέμποροι ακριβώ ε, εκμεταλλεύονται την αδυναμία ορισμένων ανθρώπων. Όσον αφορά τις ε, παράνομες υιοθεσίε, αυτό είναι κάτι που πράγματι συμβαίνει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εμπίπτει σε θέματα σωματομπορίας. Όσον αφορά την εναρμόνιση των νομοθετικών διατάξεων, ε, υπάρχουν οργανωμένες ομάδες εγκλήματος ε, και οι σωματέμποροι, οι επαγγελματίες εγκληματίες θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολύ ελκυστική αγορά να το ξαναπώ ε, μια αγορά ε, με χαμηλό κίνδυνο. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το εχθρικό περιβάλλον για αυτούς, όπως είπα, σε ορισμένα κράτη-μέλη. Είτε διότι δεν υπάρχει η σωστή νομοθεσία, είτε διότι δεν υπάρχει επαρκής ε, νομοθεσία. Διάλογος με τις ΜΚΟ. Αυτός είναι καθοριστικής σημασίας. Εγώ ασχολούμαι τη δίωξη εγκλήματος πάρα πολλά χρόνια και οι ανακρίσεις και το οργανωμένο έγκλημα είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Οι επιτυχείς έρευνες δεν μπορούν να γίνουν αποκομμένες από τις ΜΚΟ και από την κοινωνία των πολιτών. Οι υπηρεσίες δίωξης εγκλήματος δεν μπορούν ε, μόνες τους ε, να φέρουν ένα εγχείρημα σε τέλος. Ε, πρέπει να συνεργάζονται και με άλλες οργανώσεις και φορείς. Η δική μου λοιπόν η εμπειρία δείχνει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολλές αφοσιωμένες ομάδες δίωξης εγκλήματος που συνεργάζονται στενά με ΜΚΟ είτε μέσα με άτυπα μνημόνια συνεργασίες ή άτυπες συμφωνίες αλλά υπάρχει συνεργασία με τις ΜΚΟ. Η κοινωνία των πολιτών ε, πρέπει να νιώθουν εμπιστοσύνη απέναντι στου αστυνομικού, τι θα κάνουν οι αστυνομικοί με τα δεδομένα ε, και οι αστυνομικοί πρέπει και αυτοί να νιώθουν εμπιστοσύνη όσον αφορά την ανταπόκριση των θυμάτων. Το διαδίκτυο ως ε, ένα μέσο υποστήριξης της σωματεμπορίας ή ένα μέσο σωματεμπορίας. Κοιτάξτε, εξαρτάται από την εκάστοτε νομοθεσία και εξαρτάται και από την αποδοχή της επικοινωνίας, πώς ορίζεται η επικοινωνία σε κάποια χώρα. Ε, σε ορισμένες ε, επικοινωνία είναι όλα αυτά που αποστέρονται και το διαδίκτυο είναι σαφώς και εκεί, εντάσσεται και αυτό στην επικοινωνία. Το διαδίκτυο το να αντιμετωπίζει και το διαδίκτυο σε ένα μέσο ποινικοποίηση μπορείς, αυτό θα ήταν ε, μάλλον ε, εκτός πραγματικότητας. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να καταφύγουμε όσον αφορά το, έγκλημα, στο κυβερνο, το κυβερνοέγκλημα σε εμπειρογνώμονες. Και αυτό είναι ένα θέμα δίωξης εγκλήματος. Και είπα ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ε, σωματεμπορία και την διευκόλυνση της παράνομης ε, μετανάστευσης. Τα όρια είναι ρευστά. Υπάρχει όσμωση ανάμεσα σε αυτά τα δύο, τους δύο τομείς. Άρα δηλαδή ε, πρέπει κανείς ε, να είναι προσεκτικός ε, εφόσον εργάζεται στα σύνορα. Προηγουμένως η συνάδελφος μίλησε για την εκπαίδευση των υπαλλήλων της Frontex, οι οποίοι αναζητούν και διώκουν όλες τις μορφές εγκληματικότητας. Εγώ έχω συνεργαστεί με συναδέλφους σε χώρες που υπάρχει Frontex και αυτοί έχουν έτσι μια ευρεία ε, άποψη για τις απειλές που υφίστανται από τις οργανωμένες ομάδες οι οποίες είτε προσπαθούν να διευκολύνουν την ε, παράνομη μετανάστευση μεταναστών είτε το σωματομπόριο. Επαιτία. Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Αναφέρθηκε το θέμα των γονιών. Παράδειγμα, οι έρευνες ανάμεσα στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρουμανία Κυρίω για το ε, εμπόριο, παράνομο εμπόριο παιδιών των Αθήγανων Ρωμά. Και αυτό αφορά ε, στην ερώτηση που ετέθηκε από τον Βρετανό συνάδελφο σχετικά με τροτές ομάδε. Οι γονεί εμπλέκονται και αυτοί, είναι συνένοχοι στη σωματεμπορία. Παίρνουν προμήθεια ή πληρώνονται ένα συγκεκριμένο ποσό για να πουλήσουν το παιδί τους ή και οι ίδιοι γονείς πολλές φορές είναι σωματέμποροι. Μπορείτε λοιπόν να κατανοήσετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ανακριτές για να πάρουν μια κατάθεση από ένα παιδί όπου οι ίδιοι οι γονείς είναι οι δράστες. Τώρα ποιο παιδί θα καταγγείλει το γονιό του. Και ακόμα και αν υπάρχει και μια έννοια της ανεξαρτησίας σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά και στι καλύτερε των περιπτώσεων υφίσταται, ασκείται πίεση το παιδί να μην μπει την αλήθεια. Εγώ είσα μια περίπτωση, ένα κορίτσι δυνάμει θύμα και αυτό μεταφέρθηκε σε ένα ασφαλές μέρος και εκείνο το βράδυ έφυγε το παιδί από την προστασία, πήδηξε από το δεύτερο όροφο για να πάει πίσω στους, στην οικογένειά του, στους σωματέμπορους. Πώς μπορεί κανείς να χειριστεί ένα θύμα που δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί σου. Παιδιά λοιπόν, αντικείμενα σωματεμπορίας από τους ίδιους τους γονείς, αυτά είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για τις δυσκολίε που υπάρχουν σχετικά με τους υπόπτους ε, σωματεμπορίας. Όσον αφορά τώρα τη ζήτηση, δεν θέλω να μακρηγορήσω σε αυτό. Ε, το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα είναι, πολύ περίπλοκο. Αλλά το να ποινικοποιήσουμε την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, ε, τουλάχιστον κατ' εμέ, για μένα, είναι πολύ δύσκολο να αστυνομεύσει κάνει σε αυτό το χώρο. Τώρα, όσον αφορά τις αναφορές, τις εκθέσεις από τα Ηνωμένα Έθνη, ε, υπάρχουν σαφώς εκθέσεις σε πάρα πολλούς τομείς. Σημασία έχει να γίνονται οι έρευνες, οι, οι πέτοι να σύρονται στα δικαστήρια. Ε, πολλές φορές όμως οι καταδίκες ε, δεν ε, ανταποκρίνονται στα εγκλήματα Προφανώς ε, το σωματεμπόριο είναι επικερδές. Ε, το θύμα θεωρείται ιδιοκτησία και πράγματι πρέπει να αλλάξουμε το κλίμα, όμως το οικονομικό κλίμα που επικρατεί δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά τις ε, ομάδες πληθυσμού, πριν από κάποια χρόνια είχαμε ένα χάρτη που έδειχνε από πού προέρχονται κυρίω ε, τα θύματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω επειδή έχουν καταργηθεί ε, τα σύνορα με το Σέγγεν και το γεγονό ότι μπορεί κανεί απλά και μόνο να δείξει την ταυτότητά του όταν περνάει τα σύνορα, αυτό έχει διευκολύνει το σωματεμπόριο που αυξήθηκε. Τώρα δεν είναι εύκολο να πούμε τα περισσότερα θύματα έρχονται από την Α ή τη Β χώρα, την Α ή τη Β ομάδα. Πέρυσι, συγγνώμη λέει πρόεδρος πρέπει να τελειωνεται σιγά σιγά. Αφήστε το να μιλήσει λένε. Λοιπόν, έχουμε υπηκόους ε, Ηνωμένου Βασιλείου ε, που ε, εκμεταλλεύθηκαν άτομα για παράνομη εργασία. Επίσης, έχουμε γυναίκες απόφυτες πανεπιστημίου με δύο-τρεις γλώσσες που είναι αντικείμενα σωματεμπορίας. Υπάρχουν πάρα πολλά θύματα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει το γνωρίζουμε και πρέπει να ολοκληρώσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, έχετε και εσείς να πείτε κάτι ως απάντηση. Ναι, βλέπω πως έχουμε καθυστερήσει, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομη να πω ότι η Frontex εργάζεται μόνο σε θέματα που αφορούν στα σύνορα. Υπήρξε ένα σημαντικό ερώτημα, δηλαδή αν μπορούμε να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στην ε, παράνομη μετανάστευση και την ε, σωματεμπορία, διακίνηση λόγω σωματεμπορίας. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Εντάσσονται και αυτή την ε, παράνομη λάθρο μετανάστευση και μπορούμε να τους εφαρμόσουμε αυτή την αρχή αρκεί να μην ε, εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με νόμιμο τρόπο Αυτό που μας απασχολεί είναι η προστασία που μπορούν να χορηγηθεί στα θύματα σωματεμπορίας, ε, δηλαδή να λαμβάνουν κάποια άδεια παραμονής αφού ανακαλύψουμε ότι έχουν πέσει θύματα διακίνηση, σωματεμπορίας κλπ. Αυτό που έχει σημασία είναι η κατάρτιση και το σώματος σύνοριοφυλάκων προκειμένου να είναι σε θέση να εντοπίζουν το συντομότερο δυνατόν τόσο τους διακινητές όσο και τα θύματα. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Ο χρόνος είναι περιορισμένος για την εξακρίβωση των στοιχείων κάθε ατόμου και είναι δύσκολο λοιπόν να γίνεται αυτός ο εντοπισμός. Η κατάρτιση λοιπόν των φυλάκων είναι κάτι το απαραίτητο και να έχουν τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες σχετικά με την συμπεριφορά, τα χαρακτηριστικά και όταν έχουν κάποιον απέναντί τους να μπορούν να αναγνωρίζουν ότι είναι ε, θύμα σωματιμπορίας και να περάσουν σε μια φάση δεύτερης έρευνας ή ανάκλησης αν θέλετε προκειμένου να εξακριβώσουν αυτήν την υποψία. Ναι, η κατάρτιση είναι κάτι το ιδιαίτερο σημαντικό. Φυσικά οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Η Ισπανική Προεδρία έχει συμπεριλάβει αυτό στο πρόγραμμά της και ε, Frontex φροντίζει να παρέχει ειδική κατάρτιση για θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων και αυτό είναι ένα δύσκολο ζήτημα που πρέπει να ρυθμίζεται στο, <clears throat> σε ε, διαμεθοριακό επίπεδο. Να σταματήσω λοιπόν στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν όλα τα μέλη αυτού του πρώτου πάνελ. Θα περάσουμε ευθύ αμέσω στο δεύτερο πάνελ. Παρακαλώ το δεύτερο πάνελ να έρθει εδώ στο Προεδρείο. Έχουμε προσώπους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Θεμελιών Δικαιωμάτων, του ΔΟΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης.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 Ευχαριστώ. Περάσουμε τώρα στο δεύτερο πάνελ που αφορά τη σημασία της συλλογής προφοριών, πρόληψη και παρακολούθηση της ε, διακίνησης ε, και τις ε, πολιτικές σωματεμπορίας. Θα έχουμε λοιπόν την υπηρεσία θεμελιδών δικαιωμάτων με πρόσωπο τον κύριο Ιωάννη Δημητρακόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας κάνατε για συμμετοχή σε αυτό το σημαντικό σεμινάριο. Κυρίες και κύριοι, βασικός στόχος ε, της υπηρεσίας μας είναι να παρέχει ε, προστασία και στήριξη σε θέματα που μας απασχολούν. Το, η οργάνωσή μας οργανώ, ε, στάθηκε το 2007 και άρχισε να ξεκινάει, να εργάζεται συγγνώμη, με έρευνες ε, στον τομέα της διακίνησης εμπορίου. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει κάποιους δείκτες ε, που αφορούν τον εντοπισμό των θυμάτων, θύματα προστασίας, σε ό,τι αφορά τώρα την ε, διακίνηση ανθρώπων και τις σώματεμπορίες, εμείς καλύπτουμε τέσσερις τομείς. Τον εντοπισμό των θυμάτων, την προστασία των θυμάτων, την δίωξη των ε, δραστών και την πρόληψη της ε, διακίνησης. Αυτή οι δείκτε εφαρμόζονται στην έκθεσή μας για την διακίνηση παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δημοσιεύθηκε πέρυσι τον Ιούλιο ε, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω μερικά από τα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά την ε, εξακρίβωση των θυμάτων, ε, βασιζόμαστε σε έναν μηχανισμό συλλογής στοιχείων, όπως αναφέρθηκε προηγούμενο, βασίζεται σε έναν συγκεκριμένο ορισμό της διακίνησης, όπως αφορά την διακίνηση για οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση, για πλασματικούς γάμους κλπ. κλπ. Ε, έρευνά μας κατέδειξε ότι μόνο 8 κράτη-μέλη έχουν ε, ένα μηχανισμό συλλογής ε, στοιχείων ενώ, σε, ενώ τρεις άλλες χώρες αναπτύσσουν ένα παρόμοιο και ε, συλλογή στοιχείων γίνονται από την αστυνομία και από τη φυλακή. Ένα δεύτερο δείκτος αφορά τον αριθμό των, των παιδιών που έχουν εξακριβωθεί ως ε, παιδιά τα οποία έχουν πέσει θύματα διακίνησης. Αυτή η δραστηριότητα ε, επικαλύπτεται και με άλλες ε, παρέμες δραστηριότητες όπως η πορνεία, το λαθρεμπόριο κλπ. Το ενέκθεση του 2009 η Europol παρακαλεί τον μιλητή να διαβάζει λίγο πιο αργά το κείμενο, δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ε, περιπτώσεις ε, οι οποίες ε, έχουν, περιέχονται σε κάποιες εκθέσεις που έχουν δημοσιευθεί σε κράτη όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία όπου αναφέρθηκαν το 2009 66 περιπτώσεις, από το οποίο 88% ήταν γυναίκες, ενώ 26% ήταν ανήλικες. Ένας τρίτος δείκτης αφορά δείκτη για την ε, αξιολόγηση της εκπαίδευσης ε, του προσωπικού αλλά και των ε, μελών μη κυβερνικών οργανώσεων, επαγγελματικών υγείας κλπ. τέσσερα δεν, μας, δεν παρέχουν καμία κατάρτιση. Ε, τώρα, προστασία των θυμάτων. Ένας δείκτης αφορά την, ε, αφορά άμεσα τα παιδιά. Αυτός ο δείκτης ε, είναι πολύ σημαντικός ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ορισμένοι εφαρμόζουν την αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού και σε ορισμένε περιπτώσει όπω η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία βασίζονται σε κάποιε ε, νομικέ διαδικασίε. Ε, Επίση ε, υπάρχουν δείκτες που αφορούν τις διάφορες διατάξεις ειδικά με το δικαίωμα παραμονής. Αυτό άπτερ τη συνεργασία με τις αρχές, υπηρεσίες διώξης και τις δικαστικές αρχές. Αυτό όμως ενέχει τον κίνδυνο τα άτομα να, τα οποία έχουν συνεργαστεί με τις αρχές να παίζουν με τα θύματα αντιπίνων από τους διακινητές και τους σωματεμπόρους. Ε, στο ζήτημα αυτό δεν έχουμε πολλές, ε, πολλές στατιστικά στοιχεία. Τώρα σε φορά την δίωξη των δραστών, ένας δείκτης αφορά τον αριθμό των καταδικών και όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι έρευνες μας δείχνουν ότι οι στατιστικές αυτές έρχονται ε, σε συσχετίζονται με τις ε, στατιστικές που αφορούν τη λαθρεμπορία, την πορνεία κλπ. Αλλά υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι υπάρχουν ε, ε λίγες, λίγα τέτοια στοιχεία, ειδικά σε τέσσερα κράτη-μέλη, ανάμεσα στο 2000 και 2007. Ε, υπάρχουν και κάποια άλλα κράτη, πέντε τον αριθμό, που, στα οποία δεν αναφέρουν καμία καταδικαστική απόφαση. Πολύ συχνά οι συλλήψεις ε, δεν οδηγούν ε, στην δίωξη ή, τις, ε, ή σε καταδίκες. Τα πρόσφατα στοιχεία που λάβαμε δείχνουν ότι 400, στους 406 ε, 67 δεν είχαν σχέση με, την, ε, με το εμπόριο παιδί και μόνο 15 καταδικάστηκαν από 9 μήνες έως 11 χρόνια οι έρευνε ε, μα έχουν δείξει ότι σημαντικέ αλλαγέ, διαφορέ υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ενώ στην περισσότερα κράτη-μέλη υπάρχουν. Ε, ε, υπάρχει το δικαίωμα ε, έντησης στοιχεία όμως δεν έχουμε παρά μόνο για την Ολλανδία και αυτές οι αποζημιώσεις φαίνεται ότι την εξαίρεση στην πρόληψη της διακίνησης παιδιών τα αποτελέσματα με ορισμένων δικτών έδειξαν ότι τα κράτη-μέλη ε, εφάρμοσαν διάφορα στοιχεία, διάφορους δείκτες, συγγνώμη, αλλά μόνο 11 κράτη-μέλη συμμετείχαν στην, ε, στην γραμμή 116, την hotline, σε ό,τι αφορά την ε, εξαφάνιση παιδιών. Καταλήγοντας θα ήθελα να τονίσω ότι για την υπηρεσία μας η πρόταση της Κομισιόν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της ε, εμπορίας και την προστασία των θυμάτων. Ιδιαίτερα το άρθρο 7 της πρότασης αφορά, αφορά την ε, μη εφαρμογή και μη δίωξη ε, των θυμάτων θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι η σημαντικότερη πρόοδος Επίσης αυτό είναι ο τρόπος ε, για τον οποίο θα βοηθήσουμε και θα συμβάλλουμε μάλλον στην οικοδόμηση εμπιστοσύνη ανάμεσα στους θύματα και στους ε, αρχές. Τώρα τα άρθρα επίσης 10 12 14 συγγνώμη, ε, αποτελούν σημαντική πρόοδο. Ο ορισμός του σώματα στο άρθρο 2 αποτελεί σημαντική πρόοδο και θεωρούμε ότι η οδηγία θα πρέπει να περιλαμβάνει και μία αναφορά στις μορφές ε, ε, διακίνησης ε, που ιδιαίτερα πλήττει την, πλήττουν τα παιδιά. Στο πλαίσιο λοιπόν της, της συνθήκης Λισαβόνας η προτινόμενη οδηγία θα πρέπει να λάβει υπόψη και το καθεστώς των μεταναστών. Η έκθεση ΟΚΤΑ της Europol 2009 τονίζει ότι όπου εντοπίζονται θύματα υπάρχει βούληση, ε, δεν υπάρχει βούληση συνεργασίας με τις αρχές, κάτι το οποίο ακούσαμε και προλίγο. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα θύματα Ε, μπορούν να εμπιστευτούν τις αρχές και να, από την, να ξεφύγουν από την, την εξάρτηση στην οποία έχουν στην οποία έχουν περιέρθει εάν μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη απέναντι στις αρχές. Τέλος, ε, η προτινόμενη οδηγία περιέχει στο άρθρο 19 μια ρήτρα που, αναφέ, που ζητάει την Κομισιόν να υποβάλει έκθεση που θα στηρίζεται στις ε, προφορές στα όπως ε, είδαμε, συχνά δεν γίνεται κατάλληλη μεταφορά της οδηγίας, αλλά το αυτό που είναι προβληματικό είναι η εφαρμογή της. Το άρθρο 19 θα μπορούσε να ζητήσει από την Κομισιόν να λάβει υπόψη στοιχεία και προφορίες που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως επίσης για τη Europol, την Eurojust, Frontex και από άλλες ε, οργανώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ε, λάβουμε ως παράδειγμα την οδηγία για την ε, ισότητα, ειδικά το άρθρο 17, το οποίο αναφέρει ότι θα πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα κλπ. κλπ. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, and I would like uh, to give... Ευχαριστώ. Η εκπρόσωπο της Διεθνού Οργάνωση Εργασία, κυρία Μπεάτε Άντρε για το ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της εξαναγκαστικής εργασίας. Ξέρουμε ότι όλοι ότι η ΑΕΛΟ έχει κάνει μεγάλη πρόοδο σε αυτό τον τομέα. Κύριε Αντρές. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, μου κάνετε μεγάλη τιμή που με επιτρέπετε να συμμετάσχω στη συζήτηση αυτή για την προετοιμασία της σύνταξης μιας νέας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για λογαριασμό του ΔΟΕ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές του σεμιναρίου για τη δυνατότητα που μου δίνεται να παρουσιάσω τις απόψεις της ILO. Μου ζητήθηκε να δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα συλλογής πληροφοριών, πρόληψης και παρακολούθησης των πολιτικών anti-trafficking, αλλά πρώτα επιτρέψτε μου να κάνω μερικές γενικές ε, παρατηρήσεις σχετικά με την οδηγία που ε, ικανοποιεί την ILO και η ILO και άλλοι πέντε, οργα... οργανώσεις των ΗΠΑ έχουν στείλει μια κοινή επιστολή την οποία μπορείτε να βρείτε εκτός της αιθούσης. Συγχαίρουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη για τις προσπάθειες που κάνουν για να υποστηρίξουν τα θύματα τέτοιων σοβαρών εκμεταλλεύσεων. Από τότε που εγκρίθηκε η αποφάση πλαίσιο του Συμβουλίου του 2002 έχει γίνει σημαντική πρόοδο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πιο σημαντικό είναι ότι η εθνική νομοθεσία έχει προσεγγίσει και έχει ε, προσεγγίσει επίσης και τον ορισμό του πρωτοκόλου του Παλέρμο σχετικά με, την, ε, με το εμπόριο ανθρώπινων όντων. Κάτι που επιτρέπει την δίωξη και διαμεθοριακά σε όλες τις ε, χώρες μέλη και για λόγους ε, ε, εξαναγκαστικής εργασίας. Παρόλοι όμως την προσέγγιση των νομοθεσιών, ο αριθμός των διώξεων εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερος από τον αριθμό των θυμάτων. Σύμφωνα με τη συνολική εκτίμηση του ILO του 2005, τουλάχιστον 570.000 θύματα εξαναγκαστικής εργασίας υπάρχουν σε βιομηχανικές χώρες, σε βιομηχανικές χώρες και σε χώρες που ε, βρίσκονται στη κατεύθυνση της βιομηχανοποίησης ανά πάσα στιγμή, από τις οποίες 470.000 είναι θύματα ε, και ε, το 57% έχει πέσει θύμα εκμετάλλευσης και ενδεχομένως και οικονομικής και σεξουαλικής. Η περισσότερα, περισσότερα από τα θύματα αυτά είναι γυναίκες και παιδιά Υπάρχουν όμως και πολλοί άνδρες οι οποίοι πέφτουν θύματα αυτών των ε, ε, σωματεμπόρων. Θεωρούμε ότι οι διατάξεις του νέου σχεδίου οδηγίας εφόσον εγκριθούν θα βελτιώσουν τη, τη δυνατότητα διώξεων για τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι περιλαμβάνονται ελάχιστοι κανόνες για, την, ε, για τον ορισμό των εγκλημάτων και κυρώσεων στον τομέα του τράφικινγκ για παράδειγμα και ε, η συμπερίληψη της επαιτίας. Κάτι το οποίο είναι και σύμφωνο με την ε, ε, σύμβαση του ΑΕΛΟ υπαριθμών 29. Δεύτερον, το σχέδιο οδηγίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των θυμάτων και στις αποζημιώσεις. Γιατί υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στις επιτυχείς διώξεις και στην υποστήριξη που δίνονται στα βήματα, που δίνεται στα θύματα. Τρίτο, διότι οι εθνικοί εισηγητές είναι ε, σημαντικός θεσμός γιατί δίνουν ε, προτεραιότητα στην δίωξη και στην προσέγγιση των θυμάτων. Είναι σημαντικές λοιπόν αυτές οι βελτιώσεις. Παρ' όλα αυτά θέλω να τονίσω και ορισμένε ελλείψεις. Και σε αυτές ε, θα έρθω τώρα στο δεύτερο μέρος της ομιλίας μου και κυρίως για την καταναγκαστική εργασία. Παρόλη την κύρωση τη ε, σύμβαση του ILO υπαρθμών 29 σε όλες τις χώρε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πολλοί νομοθέτες ακόμη δεν έχουν αντιμετωπίσει σωστά την έννοια της, του ε, εξαναγκασμού σε εργασία και τη εκμετάλλευση. Πολύ συχνά μεταφέρουν απλώ τον ορισμό του πρωτοκόλλου του Παλέρμο χωρίς να ε, ορίζουν ειδικότερα το αδίκημα του εξαναγκασμού σε εργασία συχνά υπάρχουν και πολύ ε, άθλιες συνθήκες εργασίας και αυτό είναι βέβαια και θέμα δικαστηρίων. Η εμπειρία σε ορισμένες χώρες μέλη, ορισμένες δείχνουν ότι χωρίς την ε, συνειδητοποίηση του δικαστικού σώματος και χωρίς νέους νόμους δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχής δίωξη, αρκετά επιτυχής δίωξη δηλαδή των περιπτώσεων αυτών. Θα έρθω σε άλλες σε λίγο. Η ΑΕΛΟ χαίρεται για το άρθρο 8 του σχεδίου ε, οδηγίας που θα επιτρέψει να μην εξαρτώνται οι έρευνε και ανακρίσει από τι μαρτυρίε των θυμάτων. Η διάταξη αυτή αναγνωρίζει το γεγονό ότι πολλά θύματα μπορεί να ε, υποκύψουν σε πιέσει να αποσύρουν τι μαρτυρίε του. Εν προκειμένου, η ΕΛΟ θα ήθελε να τονίσει τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορούν να παίξουν οι επιθεωρήσει εργασία σε ορισμένε χώρες μέλη υπάρχουν περιορισμοί στις εξουσίε των ε, επιθεωρητών εργασία. Παρ' όλα αυτά οι επιθεωρητές εργασίες παίζουν σημαντικό ρόλο για τον εντοπισμό περιπτώσεων εξαναγκασμού εργασίας εκτός του χώρου της πορνεία. Αντίθετα με την αστυνομία, οι επιθεωρητές εργασία έχουν δυνατότητα να μπουν σε, οποιαδήποτε, χώρο εργασίας χωρίς ένταλμα έρευνας και μπορούν να δώσουν και πρακτικές ε, συμβουλές στους ε, εργοδότες. Οι χώρες μέλη του έλο αυτή τη στιγμή συζητούν νέα στάνταρτ για την, ε, την εργασία. Ο ΕΛΟ θα ήθελε να το λύσει επίσης μετά από τα σχόλια που έγιναν και από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ότι το βασικό καθήκον των επιθεωρήσεων εργασίας είναι η προστασία των εργαζόμενων και όχι η επιβολή των ε, νόμων περί νομοθεσίας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εκπαιδευτούν και οι επιθεωρητές εργασίας σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζόμενων για να μπορούν να προστατεύσουν τους εργαζόμενους από εκμετάλλευση. Επομένω, οι επιθεωρητές εργασία δεν είναι μόνο σημαντικοί για την πρόληψη το, του εγκλήματος της ε, ε, σωματεμπορίας αλλά και για να προσφέρουν προστασία στους εργαζόμενους. Έρχομαι τώρα στη συλλογή δεδομένων. Το νέο σχέδιο οδηγίας προτείνει την ίδρυση των εθνικών εισηγητών ή άλλων παρόμοιων μηχανισμών. Έχει δείξει εμπειρία ότι ένας ανεξάρτητος μηχανισμός ο οποίος να μην δεσμεύεται από την εντολή ενός συγκεκριμένου Υπουργείου είναι σημαντικός για να μπορεί να συλλέγει όλες τις σχετικές πληροφορίες από πλήθος πηγών. Ένα σημαντικό θέμα είναι και ο ορισμός του θύματος που έχει σχέση με το νομικό πλαίσιο που ανέφερα προηγουμένως. Το σχέδιο οδηγία προβλέπει ότι ένα πρόσωπο λαμβάνει υποστήριξη από τη στιγμή που οι αρμόδιες αρχές έχουν κάποια ένδειξη ότι ενδεχομένως το πρόσωπο αυτό να έχει πέσει θύμα ενός εγκλήματος όπως αυτό αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΔΟΕ έχει υποβάλει μια λίστα δικτών βασισμένη στην μεθοδολογία Delphi. Εμείς έχουμε εξετάσει τους δείκτες Delphi με σε ειδική προσπάθεια σε ορισμένες ε, χώρους, χώρες πιλότους και σε σχέση με επιθεωρήσεις σε νοικοκυριά. Τα αρχικά αποτελέσματα μας δείχνουν ότι 5 περίπου του ε, πληθυσμού των ε, μεταναστών εργαζόμενων που έχουν επιστρέψει είχαν οδηγηθεί σε εξαναγκαστική εργασία. Το 5% σας φαίνεται μικρό, αλλά εάν προβληθεί σε ολόκληρο τον πληθυσμό σημαίνει τελικά ένα σημαντικό αριθμό. Αυτές οι έρευνες δείχνουν ότι ένα μικρό ποσοστό όλων των προσώπων που έχουν πέσει θύματα σωματεμπορίας τελικά μπορούν να αναγνωριστούν. Ορισμένα από τα, ορισμένοι από τους δείκτες αυτούς περνούν και στις εθνικές τράπεζες δεδομένων. Εάν πρόκειται να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το άρθρο 10 θα πρέπει να υιοθετηθούν καλύτερες δομές και διαδικασίες για να μπορούν να εντοπίζονται τα ενδεχόμενα θύματα και για να συλλέγονται δεδομένα και για τα προφίλ των δραστών και των θυμάτων. Τέλος, ορισμένα σχόλια για την πρόληψη. Ο ΔΟΕ σημειώνει με ικανοποίηση ότι η προτινόμενη οδηγία απαιτεί από τις χώρες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποθαρρύνουν την ζήτηση η οποία στην ουσία οδηγεί σε όλες τις μορφές αυτές εκμετάλλευσης. Με την έννοια αυτή, ο ΑΕΡΟ θα ήθελε να ενθαρρύνει τις χώρες μέλη να επιζητήσουν κάποια συνοχή μεταξύ της προτινόμενης οδηγίας και των, και των νομοθεσιών περί απασχόλησης, μεταξύ αυτών και των διατάξεων περί ε, συμβατικής εργασίας, περί προσλήψεων και να ληφθούν υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές προδιαγραφές και διαδικασίες για την αντιμετώπιση τη σωματεμπορίας. Συχνά λειτουργούν σε διάφορες χώρες και ε, παράνομοι μηχανισμοί πρόσληψης. Τα προγράμματα που θα θεσπιστούν πρέπει να λάβουν υπόψη την ιδιαίτερη, το ιδιαίτερα ευάλωτο των γυναικών και των παιδιών. Και θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν το γεγονός ότι και οι άνδρες ε, πέφτουν θύματα ε, σωματεμπόρων για εξαναγκαστική εργασία. Ο ΕΛΟ θεωρεί την εμπλοκή των, οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών στον αγώνα κατά τη καταναγκαστική εργασία και στην εφαρμογή των προληπτικών μέτρων ω απολύτω απαραίτητο. Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για την ευαισθητοποίηση αλλά και για, την, ε, για τον εντοπισμό των θυμάτων και των δραστών στη συνεργασία με τι ε, υπηρεσίες δίωξη εγκλήματος. Και τέλο σημειώνει με ικανοποίηση ο ILO ότι το σχέδιο οδηγία έχει ένα μια έντονη προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ήθελα να τονίσω εν προκειμένου ιδιαίτερα τα άρθρα της ελευθερίας του συνεταιρίζεστε, των μη διακρίσεων των δικαιωμάτων του παιδιού και των άλλων που έχουν περιληφθεί στο επεξηγηματικό μνημόνιο. Η ε, δράση κατά της σωματεμπορίας είναι απαραίτητο να ενταχθεί μέσα σε μια συνολικότερη στρατηγική προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό είναι απαραίτητο για να καταστεί αποτελεσματική. you very much for Σας ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα να πω, εκφράσω την ελπίδα, ότι τουλάχιστον στο τέλος θα έχουμε ε, κάποιες εκτιμήσεις όσον αφορά στο μέγεθος, στην έκταση της σωματεμπορίας. Τώρα στην κυρία Λίδια Έρδη με το λόγο, πρόεδρο της ε, της Υποεπιτροπής ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, που αφορά ε, στην σωματεμπορία. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι για την πρόσκληση που έγινε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και συγχαρητήρια που προσκαλέσατε ένα πάνελ τόσο σημαντικό εργαζόμενοι πάνω στο ζήτημα αυτό πραγματικά άκουσα θέσεις που δεν είχα ακόμα υπόψη μου και ομολογώ πως ε, με εντυπωσίασε και η προηγούμενη στρογγυλή τράπεζα όπου υπόθηκε ότι ε, η εμπορία ε, ανθρώπων, ειδικά των γυναικών, δεν αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα και θεωρώ ότι ως πολιτική που είμαστε θα πρέπει να αναρωτηθούμε αναφορικά με το τι θα πρέπει να κάνουμε προκειμένου να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες όπως συνέβη με την διακίνηση ναρκωτικών. Νομίζω λοιπόν είναι πολύ πιο σημαντικό, πιο σημαντικό να πάψει να υπάρχει το εμπόριο ανθρώπων ε, από ότι το εμπόριο προϊόντων. Θεωρώ λοιπόν ότι η παρουσία μας εδώ ε, αποτελεί την απόδειξη ότι η συμφωνία η οποία συνήθω του Συμβούλου τη Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ενίσχυση τη συνεργασία ανάμεσα στα δύο όργανα μα θα πρέπει να τονιστεί και βασίζομαι σε μια ενισχυμένη συνεργασία λόγω ακριβώς ε, της θεματικής αλλά και των εμπειριών που έχουμε και η μεν και η δε. Εγώ είμαι μέλος ε, του Συμβουλίου από το 1991. Ε, εργάστηκα στην πρώτη έκθεση για την πορνεία και για την, τον εξαναγκασμό σε πορνεία και το Συμβούλιο της Ευρώπης εργάζεται από καιρό πάνω στο θέμα αυτό της εμπορίας ανθρώπων. Από το 1997 ζητήσαμε να καταρτιστεί μια σύμβαση και η σύμβαση αυτή η οποία τελικά καταψήφισε φασίστηκε στην Βαρσοβία τον ε, Μάιο του 2005. Πρόκειται για την πρώτη ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την ε, εμπορία ανθρώπων και η κοινοβουλευτική συνέλευσή μας είναι υπερήφανη για αυτό το αποτέλεσμα που αποτελεί το τέκνο της διότι η πρωτοβουλία προέρχεται από την Επιτροπή Ισότητας Ανώνων και Γυναικών αλλά και αποτελεί ένα πρώτο παράδειγμα όπου μια αντιπροσωπεία αυτής της Επιτροπής συμμετείχε στην Συντακτική Επιτροπή της Σύμβασης η σύμβαση λοιπόν αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης ετέθησε ενισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2008 και μέχρι σήμερα 28 ευρωπαϊκά κράτη, εκ των οποίων 18 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κύρωσαν τη σύμβαση και άλλες ε, υπέγραψαν και μέχρι τώρα υπάρχει μία χώρα που δεν έχει ούτε κυρώσει ούτε υπογράψει αυτήν την σύμβαση και κρίνω πως αυτό απαιτεί κάποιες εξηγήσεις. Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και πράγματι εξεπλάγει που δεν αναφέρθηκε προηγούμενα είναι ένα μέσο πολύ αποτελεσματικό σε ό,τι φορά την ε, καταπολέμηση της ε, διακίνησης ανθρώπων διότι αφορά την προστασία των θυμάτων ως πρώτη στην προτεραιότητα και όχι μόνο την δίωξη των δραστών αλλά υπάρχει επίσης και ένα ε, όργανο ελέγχου αποτελούμενο από εμπειρογνώμονες του οποίου η αποτελεσματικότητα τουλάχιστον επί χάρτου Αξίζει να μας προβληματίσει περαιτέρω αυτό το ελεγκτικό όργανο λοιπόν το οποίο αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ε, αποτελεί μια εγγύηση ανεξαρτησίας ε, της αξιολόγησης για την εφαρμογή της σύμβασης και δεν μπορώ παρά να ελπίζω πως ούτως ή άλλως όποια είναι η συνέχεια που θα προβλέπετε μέσω της οδηγίας, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης αλλά και της οδηγίας θα γίνονται ομού από κοινού διότι όχι μόνο πρόκειται για θέματα συνέπειας αλλά είναι νομίζω και κάτι το παράλογο, αν δεν μπορέσουμε να εξηγήσουμε στους ε, εκλογικό μας σώμα γιατί δύο ε, ευρωπαϊκά όργανα που δουλεύουν επί του αυτού θέματος δεν έχουν έναν κοινό μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης. Η σύμβαση να πω ότι στηρίζεται γύρω στα τρία π. πρόληψη, προστασία και διευκρινίζω πως ε, εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε όλα τα θύματα, ιδιαίτερα τις γυναίκες για τα παιδιά, αλλά και τους άντρε. φυσικά, οποιαδήποτε και είναι η μορφή της ε, εκμετάλλευσης αυτής, είτε είναι σεξουαλική, είτε καταναγκαστική εργασία, ή καταναγκασμό, καταναγκασμός σε παροχή υπηρεσιών. Και εν ώψη της ε, δωρεάς ε, και μάλλον της εμπορίας ε, οργάνων αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Ε, ε, το θέμα αυτό έδειξαν και οι πρόσωποι της Europol και της Eurojust ότι χρειάζεται η διέλευση, δεν χρειάζεται η διέλευση των συνόρων για να μπορέσει να ισχύσει ε, εμπορία σύμφωνα με την σύμβαση οι ε, διαδικασίες ε, ε, αξιολόγησης και ενοπισμού των θυμάτων είναι γνωστοί. Έχουμε ορίσει τουλάχιστον 30 μέρες, μια προθεσμία 30 ημερών και ζητάω εδώ από τους συναδέλφους του Κοινοβουλίου να διατηρήσουν αυτήν την διάταξη που ήταν πολύ δύσκολο να πετύχουμε στο Συμβουλή της Ευρώπης, διότι κανείς από τα κράτη-μέλη δεν επιθυμεί να παράσχει αυτή την ε, προθεσμία 30 ημερών στα θύματα για να μπορέσουν να αποφασίσουν πλήρη ηρεμία και νυφαλιότητα αν θέλουν να συνεργαστούν. Η παροχή ενός ε, προσωρινού, μιας προσωρινής μάλλον άδειας διαμονής ε, και εδώ να πω επίσης ότι και γι' αυτό χρειάζεται υπάρξει απόλυτη νυφαλιότητα ο πλευράς ε, θύματος. Γι' αυτό η παροχή αυτού, τη άδεια ε, διαμονής να πάρει μηχανισμή αποζημίωσης, προσφυγή και επαναπατρισμού και τα μέτρα πρόληψης ε, και προαγωγής της ισότητας ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες και να συμφωνήσω με όσα είπε η εκπρόσωπος του Διεθνής Οργάνωσης εργασίας. Είτε πρόκειται λοιπόν για ζήτημα σεξουαλικά είτε σε καταναγκασμό σε εργασία. Για τον μηχανισμό παρακολούθησης νομίζω ότι δεν χρειάζεται πλέον να, να τονίσω το οτιδήποτε μόνο το εξή. Θα σας πω ότι το ΚΡΕΤΑ ο ανεξάρτητος μηχανισμός ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης ξεκίνησε ήδη τις πρώτες ενέργειες. Δέκα χώρες ε, ε, ενέχονται σε αυτήν την παρακολούθηση, έχουν έξι, μέλη, έξι χώρες μέλη της, ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Ρουμανία και Σλοβακία και άλλες χώρες όπως η Ελβανία, η Κροατία, η Γεωργία και η Μολδαβία. Ε, οι πρώτες εκθέσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2011 και τον Οκτώβριο του 2011 ελπίζω να είναι έτοιμα τα πρώτα αποτελέσματα και ελπίζω να είναι και ικανοποιητικά αλλά και πιστικά. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να καταλήξω κάνοντας έκκληση στους εκπροσώπους των χωρών που δεν έχουν κυρώσει ακόμα τη σύμβαση να το πράξουν και στη μία χώρα η οποία ούτε υπογράψει αλλά ούτε επικυρώσει μέχρι τη στιγμή να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες διότι πιστεύω ότι αυτό είναι απαραίτητο. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας ε, και ελπίζω πως στην διάσκεψη που θα οργανώσει η Βελική Προεδρία τον Οκτώβριο και την που θέλει να οργανώσει το Συμβούλιο της Ευρώπης τον Δεκέμβριο θα βρεθούμε σε ίδιο τραπέζι για να αγωνιστούμε υπέρ των ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου και την προστασία των θυμάτων. Και αυτό είναι προς όφελος όχι μόνο των θυμάτων, αλλά και προς όφελος της ε, συνοχής, της συνέπειας. Για να φύγω όλο αυτό θα διευκολύνει και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αποτανθούμε στους, ε, στο εκλογικό μας σώμα για τις εργασίες των δύο σωμάτων μας. Ευχαριστώ. Thank you, for your uh, very interesting contribution and thank you for pointing out the necessity of... Ευχαριστούμε κυρία Έρ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση σας και για το ότι αναφερθήκατε στην εργασία ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θα ήθελα τώρα να αναφέρω κάτι αρκετά δυσάρεστο όσον αφορά την πίεση χρόνου. Αποφασίσαμε να έχουμε συζήτηση στο τέλος όλων των παρουσιάσεων. Έχουμε καταγράψει το ποιος επιθυμεί το λόγο και θα ήθελα να παρακαλέσω τους ομιλητές να παραμείνουν κοντά μας και οι συνάδελφοι να δείξουν υπομονή. Γιατί όπως βλέπετε Έχουμε θαυμάσιους ομιλητές από διάφορους ε, τομείς και θα ήταν κρίμα να μην ε, μας δοθεί η ευκαιρία να τους ακούσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τους επόμενους ομιλητές να έρθουν στο βήμα. Είναι από την ε, International Save the Children Alliance ε, από την UNICEF, ε, από την ύπατη αρμοστία προσφύγων να έρθουν στο βήμα και από την Σουηδική Αστυνομία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένουμε τώρα ε, τους επόμενους ομιλητές να έρθουν στο βήμα, όπως σας είπα. Thank you very much. I think we were quite ambitious uh, with having so many different topics. Νομίζω ήμασταν πάρα πολύ φιλόδοξοι με το να θέλουμε σήμερα το απόγευμα να θίξουμε τόσα πολλά θέματα. Νομίζω όμως ε, ότι έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και εφόσον έχουν έρθει οι συγητές θα ήθελα να τους ζητήσω να παρουσιάσουν τις ομιλήσεις και μετά στο τέλος θα γίνει η συζήτηση. Καταρχήν η Ρεμπέκα Οντάνελ από, ε, θα μας μιλήσει για την ε, ε, πολιτική σχετικά με την αίτηση ασύλου και τη μετανάστευση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω σήμερα εδώ. Ο οργανισμός Save the Children δραστηριοποιείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Διακοπή. Έχουμε λοιπόν ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην ε, σωματεμπορία παιδιών ε, και στην Ευρώπη και σε ε, διεθνές επίπεδο. Εγώ λοιπόν θέλω να σας μεταφέρω τη δική μας τη δουλειά όπως επίσης και τις ευρωπτικές που υπάρχουν. Η ομάδα μας λοιπόν έχει καταθέσει μία πρόταση σχετικά με την οδηγία και εκεί αναφέρονται οι αντιδράσεις που υπάρχουν. Ας εστιάσουμε λοιπόν την προσοχή μας σε ορισμένα θέματα που είναι πολύ σημαντικά για την είναι υποστήριξη των ατόμων που είναι θύματα σωματεμπορίας. Ας δούμε λιγάκι τι γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ακούσαμε, η σωματεμπορία σημαίνει εκμετάλλευση. Με απειλή, με βία, ε, μπορεί κανείς να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης με διάφορους τρόπους, ε, καταναγκαστική εργασία, επαιτία, σεξουαλική εκμετάλλευση. Πρόκειται λοιπόν για κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, για τα παιδιά αυτό σίγουρα προϋποθέτει αυτή τη βία. Άρα δηλαδή πρέπει όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε ε, την σωματεμπορία αλλά και να στηρίξουμε τα θύματα. Ε, προλαλήσαντες ανέφεραν τι σημαίνει η βοήθεια και η υποστήριξη συμπεριλαμβανομένης και της ε, ε, φυσικής και της ψυχολογικής υποστήριξης. Εγώ θα υπογραμμίσω τρία βασικά θέματα. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την πρόσβαση στην υποστήριξη. Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί ως δικαίωμα. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να είναι συνάρτηση του κατά πόσον επιθυμεί το θύμα να είναι μάρτυρας. Ε, γιατί όπως είπαμε τα θύματα δεν είναι πάντα σε θέση να συνεργαστούν. Δεύτερον, η πρόσβαση στην υποστήριξη και τη βοήθεια πρέπει να προσφέρεται σε όλους όσοι έχουν πέσει στα χέρια των σωματεμπόρων, τόσο από χώρες ε, εκτός Ευρωπαϊκής ε, όσο και σε άλλους. Όσον αφορά τα παιδιά, ε, χρειάζεται ειδική βοήθεια γιατί τα παιδιά αυτά πρέπει να ενταχθούν μέσα σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας παιδιών που καλύπτει τις ε, ανάγκες τους και τα δικαιώματά τους. Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές συστάσεις όπως ακούσαμε προτείνεται η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σημαντικό βήμα προς τα εμπρός σε σχέση με την απόφαση του 2004 δεν αναφέρεται μόνο στην αντιμετώπιση αλλά και στην πρόληψη ε, και στην ε, προστασία των ε, δικαιωμάτων των θυμάτων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το ότι η πρόταση καλεί τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι η βοήθεια αυτή δεν είναι συνάρτηση της προθυμίας του θύματος να λειτουργήσει ως μάρτυρας. Αυτό είναι σαφώς πρόοδος, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να εναρμονιστεί με τη διεθνή. Εκείνο όμως που δεν είναι σίγουρο είναι κατά πόσον τα άτομα που έχουν υποστεί τη σωματεμπορία από τρίτες χώρες, κατά πόσον αυτά θα βοηθηθούν με βάση την οδηγία. Οι προτάσεις δείχνουν ότι ε, η οδηγία 2004 ε, είχε ως προϋπόθεση τον τόπο κατοικίας. Αυτό πρέπει να το σκεφτεί το Κοινοβούλιο. Εδώ καλούνται τα κράτη-μέλη να εκδώσουν άτομα που παραμένουν παράνομα στην επικράτειά της. Και εδώ δεν υπάρχει εξαίρεση για όσους είναι θύματα σηματεμπορίας. Άρα δηλαδή αν δεν υπάρξουν άλλες διατάξεις, τα θύματα ε, εκδίδονται από τη χώρα ανεξάρτητα ε, και χωρίς να έχουν δεχθεί υποστήριξη. Η οδηγία του 2004 προβλέπει κάποια βραχία παραμονή αλλά περιορίζεται μόνο σε όσους συνεργάζονται σε ποινικά δικήματα. Η οδηγία του 2004 μπορεί να αναθεωρηθεί εν ευθέτω χρόνο. Όμως επειδή έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας και αυτή προβλέπει πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα προστασίας και μετανάστευσης, εμείς καλούμε το Κοινοβούλιο να σκεφτεί κατά πόσον η τρέχουσα πρόταση δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον την αναγνώριση ότι όλα τα θύματα πρέπει να την χάνουν της υποστήριξης. Αυτό είναι δικαίωμά τους ανεξάρτητα από το καθεστώς τους ε, της μετανάστευσης. Υπάρχουν ε, πολλές ε, πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν κενά. Και η προτινόμενη οδηγία με ολιστική προσέγγιση θα πρέπει να είναι το εργαλείο κλειδί για να εντοπιστούν οι βασικές αρχές έτσι ώστε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των θυμάτων. Και οι σχέσεις αυτών των ατόμων πρέπει να καταδειχθούν, ε, ας πούμε, ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη αν είναι παιδιά ή αν είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Για τα παιδιά, τα κράτη-μέλη πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για να προστατεύσουν τα παιδιά. Εκείνο που εμείς συστήνουμε είναι η οδηγία να αναγνωρίσει ότι αυτή η ειδική βοήθεια θα πρέπει να ενταχθεί μέσα σε ένα ευρύτερο σύστημα προστασίας των παιδιών. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι τα συστήματα αυτά αποτελούνται από διάφορα στοιχεία που αν συντονιστούν μπορούν να ενισχύσουν το προστατευτικό περιβάλλον γύρω από κάθε παιδί. Πολυτομιακός συντονισμός, πάρα πολλά θέματα περιλαμβάνονται εδώ. Έτσι λοιπόν η οδηγία προβλέπει ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες πρέπει να συντονίζονται με τις εθνικές υπηρεσίες ε, για τα παιδιά και να ενταχθούν ε, στα συστήματα προστασίας παιδιών. Άρα δηλαδή τα θύματα παιδιά, ε, αυτά είναι το πρώτο μας μέλημα και τα δικαιώματά τους με βάση την εθνική νομοθεσία η ειδική υποστήριξή τους ε, είναι μόνο ένα μέρος ε, της υποχρέωσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρίως σε σχέση με τις ε, τρίτες χώρες και σε σχέση με την επαιτία που ακούσαμε. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ε, διασφαλίσει κανείς ε, κατά πόσον πράγματι εδώ υπάρχει εμπορία. Το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Όταν τα παιδιά αποκόπτονται από τις οικογένειές τους, η πρόταση προβλέπει να υπάρχει ειδικό εκπρόσωπος αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Όμως δεν υπάρχει ορισμός αυτού του ειδικού εκπροσώπου και αυτό να αντικατασταθεί με έναν ανεξάρτητο ε, φύλακα προς όφελος του παιδιού υπάρχει ε, μια οδηγία σχετικά με τα συνόδευτα ανήλικα και ο ρόλος αυτός του φύλακα είναι πολύ σημαντικός. Ε, πρέπει να υπάρχουν διατάξεις για τους φύλακες αυτούς όπως προβλέπεται και στην πρόταση για την επαναπροώθηση. Εμείς θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δει κατά πόσο είναι δυνατόν να προστατευθούν τα δικαιώματα όλων των παιδιών που ζουν χωριστά από τους γονείς. Αυτά τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο παίζουν ρόλο στο να διασφαλιστεί ε, ο εντοπισμό αυτών των παιδιών, αλλά και προφυλάσσονται τα παιδιά. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία την προηγούμενη εβδομάδα το Συμβούλιο Ιστορικών Υποθέσεων κάλεσε την Κομισιόν να σκεφτεί κατά πόσον η κοινωτική νομοθεσία προσφέρει επαρκή προστασία, εγγύησης για όλα τα ασυνόδευτα παιδιά, ανεξάρτητα κατά πόσον ζητούν άσυλο, είναι θύματα σωματεμπορίας ή παράνομοι μετανάστες. Τα παιδιά αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως παιδιά καταρχήν μέχρι αποδείξει του εναντίου. Το Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να σκεφτεί κατά πόσον είναι απαραίτητο να υπάρχουν νέα ολοκληρωμένα μέτρα. Γιατί δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε. Υπάρχουν περιορισμοί στις, ε, ε, στην προστασία που προσφέρεται στα παιδιά από τρίτες χώρες. Και η προτινόμενη οδηγία δεν προσφέρει εγγυήσεις. Ε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά ε, θα σταλούν πίσω σε μια χώρα που θα πέσουν πάλι και στα χέρια των σωματεμπόρων. Ούτε η οδηγία αυτή είναι αρκετά σαφής επί του θέματος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ορισμένες χώρες σκέπτονται να οργανώσουν κέντρα στις χώρες προέλευσης όπου θα μπορούν να αποστείλουν πίσω τα παιδιά. Ακόμα και σε χώρες όπως το Αφγανιστάν που αγωνίζεται για ένα σύστημα προστασίας παιδιών. Τι είδου εγγύησει υπάρχουν στο Αφγανιστάν για να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά αυτά δεν θα γίνουν βορρά των ε, σωματεμπόρων. Το Κοινοβούλιο πρέπει να μεριμνήσει για περισσότερες ε, δικλείδες ασφαλείας και η οδηγία αυτή είναι μόνο το πρώτο βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Ε, να πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες συστάσεις, συστάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη ε, μπορούν να ενθαρρυνθούν, ε, να ε, λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Όσον αφορά την μη εφαρμογή των κυρώσεων ε, το, το άρθρο το σχετικό πρέπει να τροποποιηθεί για να προβλέπονται κυρώσεις. Και όσον αφορά το δικαίωμα της αποζημίωσης των θυμάτων εμείς προτείνουμε να υπάρξει μια πρόταση και αναθεώρηση των διατάξεων για τα θύματα εγκλημάτων έτσι ώστε τα θύματα να μπορούν να διεκδικήσουν ε, αποζημίωση και εκπροσώπηση. Ε, μπορούν να ε, ζητήσουν και άλλα μέτρα πέρα από τη δίμευση της περιουσίας σωματεμπόρου. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Εμείς λοιπόν καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει την πρόταση της Κομισιόν και επίσης να, ζητήσει, να ζητάει το Κοινοβούλιο ε, συνεχείς βελτιώσεις. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην επόμενη ομιλήτρια, στην κυρία Φαντέλα Νόβακ Άιρονς. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή σήμερα να σας μιλήσω εκ μέρου ε, έξι οργανισμών της UNHCR, της UNICEF, του Οργανισμού των Εθνών για τις γυναίκες και ε, πολλές άλλες, όπου συνεργαστήκαμε για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σωματεμπορία. Έχουμε λοιπόν μια επιστολή που καλύπτει τα βασικότερα θέματα ε, που θεωρούμε εμείς ότι έχουν σχέση με, το, με τη σωματεμπορία. Επίσης ε, προβλέπονται και συστάσεις ε, που ελπίζουμε ότι θα είναι χρήσιμες. Αυτή λοιπόν η επιστολή μας ε, θεωρούμε ότι μπορεί να είναι χρήσιμη. Σήμερα λοιπόν θα εστιάσω την προσοχή μου σε ορισμένα από τα πιο πιεστικά θέματα που περιλαμβάνονται στην απάντησή μας. Ως φορείς των Ηνωμένων Εθνών εμείς αξιολογούμε και εκτιμούμε τις προσπάθειες και τον ενδιαφέρον των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση των ατόμων ένα έγκλημα το οποίο περιλαμβάνει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων. Ε, ε, Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν θύματα τα οποία χρειάζονται την προστασία, χρειάζονται την υποστήριξη και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο εμείς καλωσορίζουμε την ε, πρόθεση αυτής της οδηγίας ε, όσον αφορά στους κοινοτικούς κανόνες και στην αντιμετώπιση της σωματεμπορίας. Βεβαίως αν δεν υπάρχει ε, ολιστική προσέγγιση, αυτό νομίζουμε ότι δεν είναι σωστό, θα πρέπει να περιλαμβάνονται αυτές οι τρεις λέξεις κλειδί που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Η οδηγία λοιπόν είναι η ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσει αυτή την ολιστική προσέγγιση και να την ενισχύσει με τον έλεγχο. Θα επανέλθω αργότερα στο θέμα του ελέγχου. Όσον αφορά τώρα την προσέγγιση των ΗΕ, πριν από λίγες ημέρες ο ειδικό εκπρόσωπος των ΗΕ για τη σωματεμπορία, η ειδική εκπρόσωπος, η κυρία Τζο Ζέιλο, υπενθύμησε ότι όλες οι προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η σωματεμπορία πρέπει να κατοχυρώνονται σε μια προσέγγιση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά την πρόταση, αυτή βέβαια επισημαίνει ότι υπάρχουν περιορισμοί. Τέτοιου είδους ε, περιορισμοί ε, αφορούν στην προστασία, η οποία προσφέρεται μόνο εφόσον υπάρχει ποινικό αδίκημα. Και εδώ γίνεται αναφορά στο άρθρο 11, παρότι ο στόχος είναι να υπάρχουν ειδικά προστατευτικά μέτρα για οποιοδήποτε θύμα σωματεμπορίας. Ελπίζουμε λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μπορέσουν να άρουν αυτούς τους ε, περιορισμούς στην ε, προστασία ε, που αναφέρονται στην οδηγία. Κυρίως θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να επαναληφθεί η θεμελιώδης αρχή της μη επαναπρόθεσης που δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη όχι μόνο με βάση τη Σύμβαση περί προσφύγων του 1951, αλλά και με βάση την Ευρωπαϊκή ε, Συνθήκη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εδώ θα ήθελα να σας παραπέμψω κυρίως στο άρθρο 19 του Ευρωπαϊκού Χάρτη για προστασία στην ε, περίπτωση έκδοσης ή απέλασης ε, κάτι που έχει αρκετά μεγάλη σημασία με τη σωματεμπορία. Το άρθρο 19 προβάλλει την αρχή της μη επαναπρόθεσης. Κανείς δηλαδή δεν μπορεί να σταλεί σε ποινική δίωξη, να ε, απελαθεί με περαιτέρω εξέλιξη την δίωξή του. Αυτή λοιπόν η οδηγία θα πρέπει να ισχύει χωρίς ε, καμία εξαίρεση και όσον αφορά στη σύμβαση του 1951. Η αξιολόγηση των αναγκών προστασίας των θυμάτων είναι εκείνη που καθορίζει κάθε φορά τα προσλήψιν μέτρα. Ανάλογα με τις συνθήκες ε, στη χώρα προέλευσης, ε, η ε, εθελοντική επιστροφή, αυτό μπορεί να είναι μια λύση, αλλά όχι και η μόνη. Η αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα και η προστασία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, είναι ένα βασικό στοιχείο προστασίας για ορισμένα θύματα. Όμως η προστασία είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν εθνικοί μηχανισμοί παραπομπής όπως συστήνει και η ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την λαθρεμπορία. Και αυτά σε συνεργασία με φορείς υποστήριξης. Εδώ θέλουμε να παραπέμψουμε στο προτινόμενο άρθρο 10 υπαριθμών 4. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός στα κράτη-μέλη. Επιπλέον, σε μία μελέτη η οποία έγινε από τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με την, τον εντοπισμό των θυμάτων σώματεμπορίας και η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2009, βλέπουμε ότι ε, λήφθησαν αρκετά μέτρα για να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα ανάμεσα στις διαδικασίες που αφορούν στα θύματα τις σωματεμπορίες και τα διεθνή συστήματα προστασίας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ενθαρρύνουμε να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις αρχές δίωξης και στις ε, ε, αρχές χορήγησης ασύλου. Όσον αφορά τώρα ε, τους εθνικούς μηχανισμούς παραπομπής, αυτοί μπορεί να είναι αποτελεσματικοί μόνο εφόσον οι τα αρμόδια στελέχη είναι εκπαιδευμένα. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς χαιρετίζουμε τις διατάξεις για την εκπαίδευση ε, του άρθρου 15, ε, κυρίως την ε, εκπαίδευση συνοριοφυλάκων, επιθεωρητών εργασίας, δικαστών και προσωπικού παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας. Είναι απαραίτητο να υπάρχει εκτεταμένη εκπαίδευση γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχουν και ε, εκτεταμένοι μηχανισμοί προστασίας. Κατά τη δική μας άποψη, το δικαίωμα στην νομική προστασία είναι καθοριστική σημασίας. Είναι καθοριστική σημασίας έτσι ώστε η προστασία να μπορεί να προσφερθεί στην πρακτική. Κυρίως εφόσον έχουμε να κάνουμε με περίπλοκες ευρωπαϊκές διαδικασίες. Τα θύματα της ε, ε, σωματεμπορίας πολύ συχνά χρειάζονται έναν νομικό σύμβουλο. Η δωρεάν, νομική, δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών είναι ένα μέτρο προς όφελος ε, των κρατών, καθότι μπορεί να βοηθήσει ε, να εντοπιστούν έγκαιρα και με σαφήνεια και ορθά οι ανάγκες ε, προστασίας. Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ στην μη δίωξη θυμάτων σώματεμπορίες που αναφέρεται ε, στο άρθρο 7. Εμείς χαιρόμεθα για το ότι συμπεριλαμβάνεται αυτή η πρόταση. Όμως ανησυχούμε σοβαρά για το ότι η προτινόμενη διάταξη αφορά μόνο τη δυνατότητα της μη δίωξης ή επιβολής ε, κυρώσεων. Και εδώ θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σωματεμπορία. Και παραθέτω, τα θύματα δεν πρέπει να ε, κρατούνται σε φυλακές ε, ή να καταδικάζονται ε, για το ότι συμμετείχαν σε παράνομες ενέργειες, καθότι αυτές οι παράνομες ενέργειες είναι άμεσα συνεπακόλουθο της ε, κατάστασής τους. Εμείς λοιπόν ζητούμε να μην ε, επιβάλλονται κυρώσεις σε θύματα σωματεμπορίες εφόσον αυτά έχουν εμπλακεί σε παράνομες δράσεις. Γιατί εξαναγκάστηκαν να το πράξουν αυτό παρά τη θέλησή τους. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος, δεν θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο θέμα της ε, νομικής βάσης και το ότι δεν γίνεται αναφορά στο άρθρο 79. Θα ήθελα απλά να σας παραπέμψω στην κοινή μας επιστολή και προχωράω στο να επισημάνω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια προσέγγιση ευαίσθητη ως προς το φύλλο. Οι περισσότερες διατάξεις ε, αναφέρονται με τον ίδιο τρόπο στους άνδρες και τις γυναίκες ε, ενώ δεν είναι αλήθεια. Είναι διαφορετικές οι εμπειρίες τους. Οι γυναίκες και τα κορίτσια υφίστανται πάρα πολύ βαριές επιπτώσεις, ενώ οι άντρες δεν βρίσκουν εύκολα πρόσβαση σε προστασία. Γι' αυτό λοιπόν μη ζητάμε να υπάρχει ισότητα των δύο φύλων και αυτό να συμπεριληφθεί στην διατύπωση και εφαρμογή προγραμμάτων. Να υπάρχει και η σωστή εκπαίδευση για όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους. Θα θέλαμε να σε ενθαρρύνουμε να υιοθετήσετε μία προσέγγιση που να αφορά ιδιαίτερα στα τροτά άτομα συμπεριλαμβάνοντας στο κείμενο την, ε, ε, την ευαισθησία ή το τροτό των θυμάτων με βάση το φύλλο. Όσον αφορά τώρα τον έλεγχο, ε, εδώ θέλω να σας πω ότι πρόκειται για μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να συμπεριλάβει στους κανόνες της μια διάταξη σχετικά με την εναρμονισμένη συλλογή δεδομένων. Και θέλω να υπογρομίσω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν και δεδομένα για την υποστήριξη των θυμάτων, ε, δεδομένα για την παραπομπή σε διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Εμείς χαιρετίζουμε την πρόταση να υπάρχουν εθνικοί εισηγητές και επιπλέον όσον αφορά τον έλεγχο και τους μηχανισμούς αναφοράς, θεωρούμε την η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επωφεληθεί από τον διορισμό ενός εισηγητή κατά της σωματεμπορίας, έτσι ώστε να υπάρχει και συνεπής προσέγγιση σε όλα τα κράτη-μέλη, με στόχο ορατές ενέργειες κατά των θυμάτων ε, κατά της σώματεμπορίας. Να υπάρχει έλεγχος και σύστημα αναφοράς στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Κυρία Πρόεδρε, δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω αν δεν αναφερόμουν ε, στο ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η προστασία που προσφέρεται στα θύματα της σωματεμπορίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως το συμφέρον του παιδιού. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν περαιτέρω διατάξεις ως προς το ε, συμφέρον του παιδιού, να αναζητηθούν ε, λύσεις διαρκείας για τα θύματα, είτε πρόκειται για την ένταξή τους ε, στην κοινωνία, είτε για την επανένωση με την οικογένειά τους. Το πρόγραμμα δράσης για ασυνόδευτους ανηλίκους προβλέπει μεγαλύτερη προστασία για θύματα παιδιά. Τελειώνω, τελειώνω. Ε, Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι απαραίτητο να υπάρχουν νομικέ διατάξει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω. Thank you very much. Uh, we are really... Σας ευχαριστούμε και εμεί πάρα πολύ. Ε, σας ευχα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λυπούμεθα πολύ ε, που υπάρχει πίεση χρόνου στους τελευταίους ομιλητές, αλλά εγώ ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε το λόγο σε όλους, να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να μιλήσουν. Ε, και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, Μάτς Πάουλσον από την Σουηδία. Και αν μπορείτε να παραμείνετε στο χρόνο που έχει προβληθεί εσάς, θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Υπέροχη, υπέροχη είναι αυτή η ευκαιρία ε, που μου δίνεται να έρθω από το Gothenburg στη Σουηδία ως αστυνομικός να σας πω ε, τι κάνουμε. Εγώ δουλεύω κυρίως βράδια και νύχτες. Μακάρι να μπορούσατε να έρθετε μαζί μας στις ε, νυχτερινές μας βάρδιες στις, στα διάφορα κλαμπ και άλλα κέντρα και να δείτε πραγματικά τι σημαίνει σωματεμπορία από κοντά όπως μου εξηγήσατε δεν έχω πολύ χρόνο. Ε, επομένως ε, θα προχωρήσω ευθύς αμέσως στην ουσία. Εφτά χρόνια τώρα ασχολούμαι με τα θέματα αυτά και είναι πραγματικά βρώμικη δουλειά από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχω πάει στο Κουρδιστάν, στο Καζακστάν, στην Μολδαβία. Ήρθαν και μας επισκέφθηκαν άνθρωποι από την Νιγηρία, από την Νορβηγία, από τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ιταλία είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με ανθρώπους από όλες τις χώρες αυτές και είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Ναι. Ε, τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε ότι αποκτάμε μία σαφή εικόνα. Έχουμε εκπροσώπους από χώρες όπου τα μικρά παιδιά ή, ή τα αγόρια είναι αντικείμενο αγοραπολισίας και ε, δυστυχώς δεν μπορούμε να δεχθούμε το ότι ε, μπορεί κανείς να αγοράζει έναν άνθρωπο απλά και μόνο επειδή έχει λεφτά ή επειδή θέλει να κάνει έρωτα σεξ με το κορίτσι. Είναι να μην μπορεί ε, να, επιθυμεί. αγοράσει κάποιο νεφρό, διότι έχει νεφρό που δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Υπάρχουν λοιπόν ε, απαγωγές ε, οι οποίες γίνονται και φυσικά πολλές φορές ε, σε αυτό συμβάλλουν και οι διεφθαρμένες αρχές. Ως ε, αστυνομικός έχω δύο στόχους στο επάγγελμά μου. Πρώτα απ' όλα να μπορέσω να ανακαλύψω τις οργανώσεις που κρύβονται πίσω από την ε, εμπορία ανθρώπων αλλά και να εντοπίσω επίσης τα θύματα αυτών των ε, δραστών και να τους προσφέρουμε μια καινούργια ζωή. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με ε, κοινωνικούς φορείς, με μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε ό,τι αφορά τις ε, οργανώσεις αυτές καταλαβαίνουμε πρέπει να στοχεύουμε τόσο υψηλά όσο και χαμηλά αφενός τους τα, τα στελέχη αλλά και τους τους χρήστες, ε, τους πελάτες, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτοί που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες ε, έχουν πέσει σήματα σώματεμπορίας. Και θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στα προγράμματα για, τους, ε, για τα άτομα τα οποία συνεργάζονται με την αστυνομία. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα Ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο ή τρεις ε, Ρωσίδες ή Νιγεριανές ε, γνωρίζουμε ότι κυκλοφορούν στους δρόμους του Γκέτεμποργκ και που εξαρτώνται από μια οργάνωση, συλλέγουμε μαρτυρίες αλλά και αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να θέσουμε τέλος στην δραστηριότητα αυτών των οργανώσεων. Έχουμε σε επαφή με κοινωνικούς φορείς, και τους ε, ενημερώνουμε για τα, για τα τις αυτές αλλά και για τα ακόρια συχνά τα οποία τις περισσότερες φορές είναι ανήλικα τους ζητάμε να ετοιμάσουν ε, κάποιους χώρους υποδοχής ε, προστατευμένους και όταν λοιπόν μπαίνουμε σε δράση τότε παίρνουμε τα άτομα αυτά τα μεταφέρουμε στους ε, κατάλληλους χώρους και τα προστατεύουμε. Ασχολούμεθα με τα θύματα, όπως καταλαβαίνετε, τα οποία και ανακρίνουμε ε, στο μικρό τμήμα, τους ζητάμε την ε, εθνικότητά τους, την ηλικία τους και για ποιο λόγο βρίσκονται στην Σουηδία, πώς έφτασαν, τι κάνουν ακριβώς. Δεν, τους, δεν τα ρωτάμε φυσικά εάν πρόκειται για εκπορνευόμενα άτομα, αν ε, παρέχουν κάποιες άλλες υπηρεσίες, ε, είναι εργατικό δυναμικό κλπ. Αυτό δεν το κάνουμε σε πρώτη φάση, διότι γνωρίζουμε πως συχνά οι απαντήσεις σε αυτή την πρώτη φάση είναι εσφαλμένες, είναι ψευδείς, ότι τους έχουν ε, πει οι οργανώσεις που τους εκμεταλλεύονται πώς θα πρέπει να απαντήσουν σε τέτοιου ερωτήσει. ερωτήσεις. Τους δίνουμε χρόνο, προσπαθούμε να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη τους, τους ε, ακούμε και σιγά σιγά αποκαθίσταται ανάμεσά μας ε, ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συχνά μεταβαίνουμε στις περιοχές αυτές του Γκόντεμπουργκ, παίρνουμε κάποιες φωτογραφίες και τους τις δίνουμε, παίρνουμε φωτογραφίες ε, από κάποια πάρκα κλπ, τις οποίες στέλνουν στους ε, γονείς του ε, για να του δείξουν ότι διασκεδάζουν, ότι παίρνουν καλά στον Κότεμπουργκ κλπ. Το εμείς όμως ε, φροντίζουμε να τους βοηθήσουμε, να έρθουν σε επαφή με τις ε, οικογένειε τους, τους παίρνουμε σε κάποια καφενεία για να πιούμε έναν καφέ κλπ. Δεν του μιλάμε καθόλου για θέματα ε, πορνείας κλπ. Διότι είναι άτομα οξυδερκοί αλλά και άτομα τα οποία η ζωή τα έχει σκληραγωγήσει. Συζητάμε λοιπόν μαζί τους ε, επί παντός αν θέλετε πιστητού εάν πρόκειται για Ρώσους ή Ρωσίδες ε, τους ε, φέρνουν σε επαφή με κάποιον ο οποίος ομιλεί τη Ρωσική, έχει μεταβεί στην Ρωσία και σιγά σιγά λοιπόν χρόνο με το χρόνο τους προσεγγίζουμε και όταν περάσουμε λοιπόν τις πρώτες δυσκολίες προχωράμε. Μερικές φορές ε, ε τυχαίνει να απελπιζόμεθα, αλλά αυτό δεν είναι σωστό, διότι αυτή η προσπάθεια είναι προσπάθεια η οποία θα πρέπει να διαρκέσει χρονικά. Λοιπόν, κάνουμε επίσης και κάποιες συζητήσεις τυπικού χαρακτήρα υπήρχαν 18 ε, Ρώσοι και μέσω μιας ε, γυναίκας Ρωσίδας η οποία ε, μιλούσε άσκημα σουηδικά φροντίσαμε να έρθουμε σε επαφή με τα άτομα αυτά και μαθαίναμε κάποιες πληροφορίες και έστω και τηλεφωνικά μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Μερικές φορές υποχρηνόμεθα ότι ήμασταν υποψήφοι πελάτες και ρωτούσαμε πληροφορίες σχετικά πότε θα μπορούμε να δούμε την κοπέλα, ε, αν ε, μπορώ να κάνω μαζί της το οτιδήποτε κλπ. Λοιπόν, και είναι προφανές ότι όταν ε, γίνονται τέτοιου είδου ε, συνομιλίες κατανοεί κανείς ότι πρόκειται για αγορά σεξουαλικών ε, ερωτικών υπηρεσιών. Και εμείς ε, έχοντας μαγνητοφωνήσει κάποιες συνδιαλέξεις αυτού του είδους χρησιμοποιούμε αυτές τις συνομιλίες ως αποδεικτικό στοιχείο στον δικαστήριο και αυτό φυσικά μας βοηθάει. Νομίζω πως ε, έχω μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προσωρινές άδειες ε, παραμονής, αυτό χρησιμεύει για να βοηθήσουμε τα θύματα. Συχνά πρόκειται για ε, άδειες διαμονής τριών ή έξι μηνών. Δίνει το χρόνο στα θύματα να σκεφτούν πλήρη ηρεμία και νυφαλιότητα τους δίνουμε λίγα χρήματα, όχι πολλά, λίγα, κάτι το οποίο όμως επιτρέπει να αγοράσουν μερικά είδη πρώτης ανάγκης, τους παρέχουμε φυσικά στέγη, δεν είναι τελικά πάρα πολλά αυτά, αλλά αυτά προσφέρει κοινωνική πρόνοια, διότι υπάρχουν από το σύνδρομο της Στοχόλμης, όπως λέγεται, διότι για ένα αρχικό διάστημα ε, συνεχίζουν να προστατεύουν τον προαγωγό τους ε, ή τον δημιό τους αν θέλετε πείτε το όπως ε, νομίζετε και νωρίτερα ακούσαμε ότι συχνά δεν κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε κάποιο, κάποιο οργάνωση, κάποιο κλίμα το οποίο αποτρέπει τις εγκληματικές οργανώσεις αλλά συχνά ακούσαμε, ε, συγγνώμη για την έκφραση, να το πω αγγλικά, fuck the police, fuck the Swedish law από τα άτομα αυτό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ε, θα πρέπει να πλήξουμε και τους ε, επικεφαλής των οργανώσεων αλλά και τους πελάτες. Νομίζω ότι όλες ε, θα συμφωνήσουμε ότι όντως θα ήταν πολύ χρήσιμο να κάνουμε μια νυχτερινή βάρδια μαζί σας στους δρόμους του Γκέτεμπορκ και να παρακολουθήσουμε πώς δράτε. Μαθαίνει κανείς πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ακόμα δύο συναδέλφους που ε, θα συμμετάσχουν σε συμπεράσματα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και από τον ΟΑΣΕ. Μιλώ για τα πρόσωπα Κούνο Τάρφουσερ και Μαρία Γκράτσα Τζαν Μαρίνο. Yeah, yeah. You want to organize hmm? It's okay. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ που προσήλθατε στα έδρανα του Προεδρείου δύο ε, συμπερασματικές ας πούμε τοποθετήσεις και μετά ελπίζω θα έχουμε λίγα λεπτά για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ε, σύντομη συζήτηση. Κύριε Κούνο Τάφουσερ, δικαστής των προδικαστικών τμήματων, ε, πέστε μας τα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ πρώτα για την πρόσκληση στο σεμινάριο παρόλο που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και το καταστατικό του δεν αναφέρονται στα διάφορα μέσα και μηχανισμούς του προημίου του ψηφίσματος της 10 Φεβρουαρίου 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. παρόλα αυτά θα αρχίσω να ε, αναλύοντας λίγο το νομικό κείμενο του ε, Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με το έγκλημα της σωματεμπορίας. Το θέμα, εάν δηλαδή εμπίπτει το έγκλημα της σωματεμπορίας στο καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δεν είναι τόσο απλό όσο θα ανέμενε κανείς. Από τη μια μεριά, αυτή η σωματεμπορία, καθ' αυτήν, δεν περιλαμβάνεται ως έγκλημα στο καταστατικό του ε, Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Εάν εξετάσετε τον κατάλογο των ε, δραστηριοτήτων ή των ενεργειών που μπορεί να θεωρηθούν ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μόνο πράξεις οι οποίες είναι συγγενείς με, αλλά δεν είναι ε, σωματεμπορία, μπορούν να ληφθούν υπόψη. Το άρθρο ΣΕ, για παράδειγμα, προβλέπει την ε, ε, ε, εισαγωγή σε δουλεία. Επίσης, την γενετήσια, το γενετήσιο εξαναγκασμό σε δουλεία στο G και επίσης το 7K, το οποίο ως γενική ρήτρα περιλαμβάνει στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας η αδίποτε άλλη πράξη παρόμοιου χαρακτήρα που από πρόθεση προκαλεί σοβαρή βλάβη ή τραυματισμό ψυχολογικό ή σωματικό. Επομένως, χαρακτηρίζεται η πράξη εκ των αποτελεσμάτων της. Από την άλλη μεριά, βέβαια, η σωματεμπορία, δηλαδή το εμπόριο ανθρώπινων όντων, περιλαμβάνεται στο άρθρο 7 του καταστατικού του δικαστηρίου, όπου η παράγραφος 2 περιλαμβάνει ορισμένες διευκρινήσεις σχετικά με την έννοια και το εύρος εφαρμογής των όσων διαλαμβάνονται στην πρώτη παράγραφο και ιδίω το άρθρο 7 2 γάμα ε, διαλαμβάνει και την, ε, τα περιεχόμενα της συνθήκης του 1976 και λέει ότι εισαγωγή σε δουλεία σημαίνει την άσκηση οσδήποτε ή όλων των εξουσιών που έχουν σχέση με το δικαίωμα της ε, ιδιοκτησίας επί ενός προσώπου και περιλαμβάνει και την άσκηση τέτοιας εξουσίας στην διάρκεια σωματεμπορίας και ιδίως σε βάρος γυναικών και παιδιών. Αυτά έχουν το νόημα ότι βοηθούν το δικαστήριο στην ερμηνεία του καταστατικού. Και λέει παρακάτω ότι για το λεγόμενο enslavement, την υπαγωγή σε δουλεία δηλαδή, για να, για να μπορέσει να χαρακτηριστεί έτσι μια πράξη, πρέπει ο δράστης να ασκεί κάποια εξουσία εξ όσων συναπαρτίζουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί προσώπου όπως για παράδειγμα την πώληση ή ε, ανταλλαγή προσώπου που συνεπάγεται βέβαια την στέρηση της ελευθερίας του προσώπου αυτού. Τέλος της παράθεσης. Υπάρχει και μια υποσημείωση που περιλαμβάνει μια εξήγηση με τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος και νομίζω ότι οι συντάκτες των ορισμών αυτών ίσως δεν είχαν τόση εμπιστοσύνη στην κρίση των δικαστών, διότι υπάρχουν τα άρθρα και υπάρχουν τα υποπαράγραφοι και υποσημειώσεις. Όλες αυτές και λέει ότι ε, θεωρείται ότι εν προκειμένου περιλαμβάνεται και η σωματεμπορία και κυρίως σε βάρος γυναικών και παιδιών. Η ίδια διατύπωση περιλαμβάνεται και στο τμήμα ε, χαρακτηριστικά στοιχεία εγκλημάτων. Θα πρέπει να προσθέσω ωστόσο ότι η από τις συμπεριφορές που αναφέρονται στο άρθρο 7 και που σημαίνουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μόνο όταν ασκούνται ως τμήμα συστηματικής επίθεση κατά ιεσδήποτε πληθυσμιακή ομάδα εν γνώση της επίθεσης. Αυτό αποτελεί και το πλαίσιο για την άσκηση τέτοιων εγκλημάτων κατά τη ανθρωπότητα. Τώρα, η συμπληρωματικότητα. Όσα αυτά, όλα τα στοιχεία αυτά που αναφέρονται στην ε, σωματεμπορία διαφέρουν κατά το ότι κατά το πώς μάλλον διαμορφώνουν τη σχέση μεταξύ των δύο. Δηλαδή, το καταστατικό θεωρεί το trafficking ως μία από τις συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε σκλαβιά. Τα international instruments μιλούν για την εισαγωγή σε σκλαβιά ως ένα από τα στοιχεία που μπορούν να αποτελούν την σωματεμπορία. Δηλαδή, η σωματεμπορία είναι στενότερη ως από την, εισαγωγή από την υπαγωγή σε σκλαβιά μάλλον. Υπάρχει μια μερική επικάλυψη βέβαια που ίσως όμως να έχει κάποια ε, συνέπεια στην άσκηση ε, δικαιοδοσίας στο εθνικό και διεθνές επίπεδο εδώ. Ως γνωρίζετε η άσκηση δικαιοδοσίας από πλευράς του δικαστηρίου κυριαρχείται από το στοιχείο την αρχή της συμπληρωματικότητας. Υπάρχει δηλαδή καταρχήν υποχρέωση των χωρών να ερευνούν τα εγκλήματα αυτά και το Διεθνές, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παρεμβαίνει μόνο όταν η χώρα όπου θα έπρεπε να διεξαγάγει τις ανακρίσεις είναι απρόθυμη ή ανίκανη να το πράξει. Εάν η υπόθεση έχει σχέση με ε, εμπίπτει μάλλον στον στενότερο ορισμό του, της υπαγωγής σε σκλαβιά, το Διεθνές Δικαστήριο θα είχε αρμοδιότητα, θα είχε δικαιοδοσία και θα ε, ε, εφαρμόζονταν η αρχή της η κανόνες συμπληρωματικότητας. Αν όμως άλλη συμπεριφορά εκτός από την υπαγωγή σε σκλαβιά που θα, ήταν, θα σήμαινε όμως σωματεμπορία Εδώ το ερώτημα βέβαια είναι περισσότερο ακαδημαϊκού χαρακτήρα, διότι στην πραγματικότητα οι δύο ε, ορισμοί μου φαίνεται ότι συμπίπτουν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μπορούν να ε, ισχύσουν δύο προσεγγίσεις. Αφενός μπορεί να πει κανείς ότι η σωματεμπορία όπως, όπως προβλέπεται στην, ε, στο καταστατικό είναι σε γενικούς, ορισμούς, σε γενικούς όρους και μια στενότερη σε μια στενότερη ερμηνεία οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν εντάσσεται στο καταστατικό θα ήταν και εκτός της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Το συμπέρασμα αυτό το υποστηρίζει και η αρχή της, στενή, της στενής ερμηνείας των διατάξεων. Δεν θα ήταν σωστό για μένα να ταχθώ τώρα υπέρ του ενός ή του άλλου επιχειρήματος. Αρκεί να πω ότι όποια και αν είναι η προσέγγιση που θα επιλεχθεί, πάντως δεν είναι αμφιλεγόμενο ότι τουλάχιστον μία διάταξη στο καταστατικό ζητεί συνεργασία μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και σε θέματα που έχουν σχέση με τη σωματεμπορία. Και μιλώ για το άρθρο 93 παράγραφος 10 που προβλέπει ότι το, διεθνικό, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, εάν του ζητηθεί, μπορεί να, χωρί, να ε, προσφέρει τη συνεργασία του σε χώρες όχι μόνο για εγκλήματα τα οποία εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του και όπου γίνονται έρευνες στο εθνικό επίπεδο, αλλά και για συμπεριφορές, πράξεις, οι οποίες γενικά υπάγονται στα σοβαρά δικήματα υπό την εθνική νομοθεσία της συγκεκριμένη χώρας. Και επειδή δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σωματεμπορία ανθρώπινων όντων είτε περιλαμβάνεται είτε όχι στην ερμηνεία του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Πάντως χαρακτηρίζεται ως βαρύ έγκλημα. Μου φαίνεται προφανές ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εντάσσεται πλέον στο σύνολο εκείνων των μηχανισμών που θα βρεθούν την πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της σύγχρονης αυτής μάστιγας. Έτσι λοιπόν στα μάτια μου αναφορά στο δικαστήριο και στο προήμιο των διαφόρων διεθνών εγγράφων που έχουν σχέση με την ε, εμπορία ανθρώπινων όντων σίγουρα θα είχε τη δικαιολογία της. Όπως έμαθα δηλαδή σε 25 χρόνια ε, υπηρεσία μου στην Ιταλία, παρόλο το όνομά μου, η συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμών είναι θεμελιώδου σημασία για να υπάρξει πραγματικά αποτελεσματικό αγώνα κατά ουδήποτε εγκλήματο. Ευχαριστώ πολύ. Μια τελευταία τοποθέτηση, συμπερασματική τοποθέτηση της κυρίας Τζαμαρινάρο του ΟΑΣΕ του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη κυρίε και κύριοι. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και την Επιτροπή ΚΑΜ που μου προσφέρουν αυτή την ευκαιρία να συμβάλλω σε αυτό το σημαντικό σεμινάριο. Να σας πω μερικά λόγια τώρα αναφορικά με την εντολή μου. Είμαι ειδικό εκπρόσωπος για την διακίνηση ανθρωπίνων όντων που ιδρύθηκε το 1993. Έχουμε ως στόχο να καταπολεμήσουμε αυτή την σύγχρονη μορφή σλόβε σκλαβιάς η εντολή μου καλύπτει και τις τρεις πτυχές των δράσεων ε, πολιτικό, θεωρητικό και ανθρώπινη διάσταση αλλά ασχολούμαι ιδιαίτερα με το ε, θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της σώματεμπορίας. Δίνουμε σύμβουλες ε, και τεχνική αρρωγή για την εφαρμογή αυτής της ε, anti-trafficking policy. Θα ήθελα να τονίσω επίσης το γεγονός ε, ότι συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς, ε, μη κυβερνικέ οργανώσεις. Την προσεχή εβδομάδα θα έχουμε οργανώσει μια διάσκεψη την οποία θα θίξουμε το ζήτημα της ε, σκλαβιάς, ε, της δουλείας, ε. και στο εγγύς μέλλον είμαι αποφασισμένη να εστιάσω ιδιαίτερα στο θέμα της εμπορίας για λόγους εργασίας και για έχει εξεταστεί ιδιαίτερο θέμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, αλλά όχι το θέμα της καταναγκαστικής εργασίας και της εκμετάλλευσης. Ε, μπορούμε να σκεφτούμε εδώ το θέμα των οικοδομών, της επεξεργασίας της τροφίμων, της αλληλείας, της γεωργίας. Κατανοούμε λοιπόν πως ε, το, ότι η εμπορία είναι μαζικό φαινόμενο, περισσότερο από ότι πιστεύαμε πριν από μερικά χρόνια. Και θα ήθελα να πω πρώτον ότι είναι αναμφισβήτητο πως πολλές προσπάθειες έχει καταβάλει η διεθνή κοινότητα, οι κυβερνήσει ε, για να αντιμετωπίσουν την εμπορία ανθρώπων, αλλά η ε, αλλά ε, το φαινόμενο είναι τεραστίων διαστάσεων και δεν έχουμε μπορέσει ακόμα να ανταποκριθούμε στο έργο αυτό. Έχουμε όλο και περισσότερα θύματα και φροντίζουμε να ε, πετύχουμε την ε, συλλήψη καταδίκη πολλών διακινητών. Η διακίνηση ανθρώπων ε, είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα αλλά και ιδιαίτερα προσοδοφόρο σε σχέση με άλλες μορφές ε, εγκλημάτων. Και έχουμε στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργάνου της Εργασίας αυτές, αυτή η διακίνηση εμπορίων ανθρώπων ε, προωθεί και ευνοεί την ε, άλλες μορφές λαθρεμπορίου όπως όπλων, ναρκωτικών κλπ. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο διονγκώνει τώρα και περισσότερο, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως είπε ο Χάρβεϊ. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πιο εχθρικό κλίμα και περιβάλλον για τους ε, διακινητές, τους δράστες και ένα πολύ πιο ευνοϊκό και φοιτικό για τα θύματα τα δύο αυτά ζητήματα είναι άρρηκτα δεμένα Τώρα η προστασία των θυμάτων ε, εμπορίας ε, είναι επιτακτικό, αλλά οι πρακτικές που εφαρμόζονται δείχνουν πως ε, είναι και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να υπενθυμίσω ότι είπε από τη Σουηδική Αστυνομία αναφορικά με τη διαδικασία οικοδόμησης εμπιστοσύνη. κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε τα θύματα. Αυτό οπωσδήποτε απαιτεί μια ικανή πολιτική, εκπαίδευση για, τους, ε, για τις αστυνομικές αρχές, στενή συνεργασία ανάμεσα στις ε, υπηρεσίες δίωξης ε, εγκλήματος ε, και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων να πω ότι είναι κάτι το οποίο είναι ευπρόσδεκτο και περιέχει κάποιες καινοτόμες προτάσεις ε, και σε σχέση με, τις, ε, με τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και να επενθυμίσω πως ε, μία από τις, μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες της οδηγίας είναι το γεγονός ότι το θύμα θα πρέπει να προστατεύεται άμεσα, δηλαδή σημαίνει ότι θα πρέπει να τύχει στήριξης ε, ακόμα και όταν ε, κρίνουμε πως ε, είναι ένα πιθανό, ένα ενδυνάμει σήμα Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συχνά μια απόφαση των αρμοδίων αρχών απαιτείται προκειμένου να ξεκινήσει η παροχή στήριξης ε, και βοήθειας ε, στο θύμα. Αυτή λοιπόν η πολιτική η προστασία θα πρέπει να μπορεί να, τεθείς, να τίθεται σε ενέργεια σε κάθε περίπτωση Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται κατάλληλοι επιθεωρητέ εργασία ε, που μπορούν να εντοπίζουν ε, εν δυνάμει τέτοιες περιπτώσεις ε, εμπορίας ή εκμετάλλευσης αλλά εν πάση περιπτώσει σε κάθε, σε κάθε περίπτωση που έχουμε λαθρομετανάστες, ε, παρανόμους εργαζόμενους. Μία σημαντική διάταξη της οδηγίας είναι αυτή που αφορά την ε, παροχή βοήθειας ε, άνευ όρων ε, υπό οποιοσδήποτε προϋποθέσεις. Ε, όταν υπάρχει λοιπόν μια υπόνοια ότι το άτομο είναι θύμα, τότε η βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται ευθύς εξ αρχής και άνευ όρων. Από το κείμενο το οποίο δημοσίευσε χθε το Συμβούλιο, βλέπουμε πως εισαγάγει κάποιους εξεχωτικούς περιορισμούς σε ό,τι φορά αυτή την αρχή της unconditional assistance και κάνω έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να βελτιωθεί το σημείο αυτό και να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την ε, προστασία άνευ όρων δίχως περαιτέρω περιορισμών. Επίσης να αναφερθώ και σε άλλα δύο ζητήματα. τα οποία η συμβολή του Κοινοβουλίου μπορεί να είναι πολύ σημαντική μετά από τη δήλωση του Συμβουλίου. Η ε, ετεροδικία είναι σαφές ότι η εμπορία ανθρώπων αναλαμβάνεται από εγκληματικές οργανώσεις που δεν είναι παραδοσιακές εγκληματικές οργανώσεις που είναι βαθιά ριζωμένες σε κάποιες ε, περιοχές όπως π.χ. ο νότος της Ιταλίας, η Δεμαθία. Υπάρχουν ε, άλλες εγκληματικές οργανώσεις που είναι εγκατεστημένες ε, στις χώρες ε, προορισμού και όχι καταγωγής θα πρέπει τα κράτη-μέλη λοιπόν να αναλάβουν την ευθύνη προκειμένου να δικάσουν αυτούς τους αλλοδαπούς εγκληματίες που έχουν ε, εγκαταστήσει το κέντρο δραστηριοτήτων τους σε ξένη χώρα. Άρα λοιπόν η ιατροδικία θα πρέπει να είναι δεσμευτική όχι μόνο για τους υπηκόους αλλά και για αλλοδαπούς. Το τρίτο θα ήθελα να τονίσω είναι το θέμα της ε, νομικής εκπροσώπησης και της νομικής αρρωγής. Ένα το θύμα μάλλον θα πρέπει να λαμβάνει μια απόφαση αφού προηγούμενα θα έχει ενημερωθεί για τις ε, δικαστικές διαδικασίες ε, και τις δυνατότητες ε, υποβολής αιτήματος αποζημίωσης. Ε, η νομική αρρωγή θα είναι δωρεάν και θα πρέπει να διασφαλίζεται ιδιαίτερα στα παιδιά και στους ανήλικους. Κάποιος είπε, νομίζω η Σίλβια Κώστα, πως ε, Ελπίζουμε πως και η οδηγία, για την, οδηγία 81 για την, του 2004 για την άδεια παραμονής ε, σύντομα θα αναθεωρηθεί. Είναι γεγονός όπως τόνισαν διάφοροι αγορητές πως ε, τα θύματα δεν είναι πάντα σε θέση να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες δίωξης του εγκλήματος και η άδεια διαμονής χορηγείται σύμφωνα με την οδηγία με βάση την ε, αρχή της συνεργασίας. Αυτό λοιπόν μπορεί να προκαλέσει εμπόδιο για μια αποτελεσματική πολιτική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί αυτό το ζήτημα και σε ό,τι αφορά τα θέματα μετανάστευσης. Να τονίσω επίσης ε, το ζήτημα των μηχανισμών παρακολούθησης. Ως ε, ΑΣΕ αναπτύξαμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά ζητήματα που αφορούν την ε, οικοδόμηση θεσμών και προωθούμε περαιτέρω αυτή τη διαδικασία. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία υπόθηκαν σχετικά με το θέμα της προτεραιότητας που πρέπει να την χάνουν τα δικαιώματα των παιδιών και της προστασίας τους. με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφορικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους, τα οποία συμμεριζόμαστε και να πω ότι η καθημερινή πρακτική θα πρέπει να αλλάξει και σε αυτό τον ζήτημα δεν θα πρέπει θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού με έναν ανεξάρτητο εκπρόσωπο του παιδιού προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση ε, και ένα συνόντευτο ε, παιδί ή ένα παιδί το οποίο έχει χωριστεί από την οικογένειά του θα πρέπει να προστατεύεται αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Thank you very much. I Σας ευχαριστώ. Η πραγματικότητα είναι βέβαια ότι δεν έχουμε χρόνο για συζήτηση. Θα προτείνουμε όμως τα μέλη των δύο επιτροπών να θέσουν ερωτήσεις και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τις διαβιβάσουμε στους ομιλητές μας και να τους παρακαλέσουμε να δώσουν άλλη φορά απαντήσεις γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε μέσα στα λίγα λεπτά που μένουν. Είμαι βεβαία ότι έχουμε πολλές ερωτήσεις. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Θα ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι όλους τους προσκεκλημένους. Έχουμε λίγα λεπτά ε, τα οποία θα καταναλώσει η Edith Bauer που είναι συνηγήτρια προσπάθησε κάπως edit να ολοκληρώσει τη συζήτηση μετά από αυτή την πλούσια ανταλλαγή απόψε. Ευχαριστώ. Έχω πραγματικά ένα μακροσκελή κατάλογο για τα όσα θα ήθελα να πω. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους που ε, με υπομονή παρέμειναν μέχρι τέλους. Βεβαίως τους ε, παρεμβαίνοντες αρχικά είχαμε προγραμματίσει 3,5 ώρες και ήμασταν σίγουρε ότι ήταν επαρκής ο χρόνος και μάλιστα και υπερβολικά πολύ. Αλλά νομίζω ότι όλοι έχουμε την εντύπωση εν τέλει ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερο χρόνο. Ε, έχουμε ακόμα πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Βέβαια δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι πάντως σαφές ότι έχουμε πολλές ερωτήσεις, περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Ένα πράγμα πάντως νομίζω γίνεται σαφές για όλες και όλους, ότι οι ευθύνες μας είναι μεγάλες, ότι πρέπει ε, η ευθύνη μας είναι μάλλον μεγάλη, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Η κύριε Λιτέρ μίλησε για την σύμβαση του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε πολλές νομικές βάσεις και χάρη στην συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και εκεί υπάρχουν ε, εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερπηδηθούν και στην έκθεση της Κομισιόν, στην πρόταση μάλλον της Κομισιόν, η οποία περιλαμβάνει ορισμένα τμήματα, αλλά ελείπουν, δεν ε, βρίσκω να είναι αρκετά ώστε να διασφαλίσουν την πρόληψη, την προστασία των θυμάτων. Ε, η πρόταση αυτή περιορίζεται σε ορισμένα, σε ορισμένα θέματα. Υπάρχουν βέβαια και καθήκοντα τα οποία ε, ξεφεύγουν από το νομοθετικό έργο και αυτά τα είπε και ο Στίβ Χάρβεϊ. Όταν κάποιο θέλει να κάνει επισκευέ στο σπίτι του αλλά θέλει να πληρώσει όσο γίνεται λιγότερα, εν τέλει αποδέχεται και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν εργάτε οι οποίοι ε, έχουν, ε, είναι θύματα σωματεμπορίας για λόγους αναγκαστικής εργασίας. Είναι ευθύνη όλων μας να πράξουμε πάντο δυνατό για να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε. ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί να κάνουμε την προσπάθεια αυτή με αποτελεσματικό τρόπο η ανοχή απέναντι στη σωματεμπορία πρέπει να μειωθεί, να μην υπάρχει. Συχνά δεν το βλέπουμε αυτό. Εμείς οι συνεισηγήτριες για το, για, το, για το νομοθέτημα αυτό πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ευαισθητοποιήσουμε τους συναδέλφους μας και βεβαίως το κοινό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ε, προσοχή σας.